Dear colleagues, uh, Αγαπητοί συνάδελφοι, πρωτού προχωρήσουμε στις ψηφοφορίες, θα ήθελα να δώσω το λόγο May I give the floor to Mr. Cavada? Στον κύριο Καβαντά. Merci, Monsieur le Président. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι. Καταρχάς, θέλω να ευχαριστήσω θερμότατα τους ε, σκιώδεις και τους ε, συντάκτες των γνωμοδοτήσεων για την εργασία που κάναμε. Κάναμε πολλές συνεδριάσεις για να προσεγγιστούν οι απόψεις με πολύ θετικό τρόπο και καταλήξαμε σε 39 συμβιβαστικέ τροπολογίε επί των οποίων συμφωνούμε. Χαίρομαι λοιπόν που μπορούμε να περάσουμε στην ψηφοφορία αυτού του αντικειμενικού, ε, συνεπούς και ολοκληρωμένου κειμένου που περιέχει τις γνωμοδοτήσεις ε, των επιτροπών των οποίων ζητήθηκε η γνωμοδότηση. Μερικά τεχνικά θέματα τώρα παρακαλώ. Στη σελίδα 2 του καταλόγου ψηφοφοριών η παράγραφος ΙΜΚΟ 25 καλύπτεται από, το συμβασμό, από τη συμβαστική πρόταση 3 και όχι όπως λέγεται τη συμβαστική πρόταση 1. Επαναλαμβάνω, η ΙΜΚΟ 25 καλύπτεται από τη συμβαστική 3 και όχι 1. Δεύτερον, στη σελίδα 7 η παράγραφος ΠΟΥΝΤ 33 καλύπτεται από τη συμβαστική πρόταση 10 η παράγραφος Κιούλτ 33 καλύπτεται από τη συμβαστική 10. Στη σελίδα 17 η παράγραφος Κιούλτ 18 καλύπτεται από τη συμβαστική 30. Στην παράγραφο, ε, η παράγραφος Κιούλτ 18 καλύπτεται από τη συμβαστική 30. Τέλος, η συνάδελφος Ρέντα απέσυρε την τροπολογία 143 αυτό σημαίνει ότι απαλήφεται η τελευταία παράγραφος της συμβαστικής 31 και αναφέρω συμβαστική 37 από εκεί που λέει η νομική θεωρητική ε, αντίληψη μέχρι παροχός legal fiction μέχρι provider στην 37 νομίζω τώρα μπορούμε να ψηφίσουμε και ευχαριστώ πάρα πολύ για την εργασία αυτή. Ευχαριστώ. Άρα εμέσως καταλαβαίνετε ότι ψηφίζουμε για την διασυνοριακή φορητότητα. Συμβαστική 1. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 165. Υπέρ. Κατά. Α, ηλεκτρονικός έλεγχος. Yeah. So, it has been adopted. Εγκρίνεται.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 Εγκρίνεται. 198 υπέρ. Α, καταπίπτει. Α, με συγχωρείτε. Συμβαστική 7 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 199 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 8 υπέρ. Συγγνώμη. Να ελέγξουμε την 199. Εγκρίνεται. Συμβαστική 8 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 202 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 33 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 206 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβαστική 9 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 33 όχι, ωραία, ναι. Συμβαστική 10 υπέρ κατά αποχέ, εγκρίνεται. 36 υπέρ κατά να ελέγξουμε παρακαλώ εγκρίνεται 35 υπέρ Α, καταπίπτει, με συγχωρείτε. 2.20 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική 11 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Ήμκο 33 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 2.28 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 38 Συγγνώμη, συγγνώμη. Πηγαίνουμε στην ΙΜΚΟ 35 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται Συμβαστική 13 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 2.37 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 40 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβαστική 14 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 2.41 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 39 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 33 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 39 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 34 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 41 και οι υπόλοιπες υπέρ κατά να ελέγξουμε παρακαλώ Απορρίπτεται. Τριάντα πέντε υπέρ κατά να ελέγξουμε παρακαλώ και εδώ εγκρίνεται 2.43 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 42 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 43 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 1 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται πιστεύω αλλά στο ελέγξουμε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 κατά αποχές απορρίπτεται 8 ε, υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 21 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 22 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 23 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 7 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 9 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 24 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 83 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 11 υπέρ κατά νοποχές ας ελέγξουμε It has been rejected. Απορρίπτεται. 25 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 91 υπέρ αποχές απορρίπτεται 26 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 27 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 14 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 28 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 29 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 115 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 15 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 17 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται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 αποχές απορρίπτεται 21 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 18 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 34 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 19 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 136 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 22 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 34α υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 21 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 35 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 24 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 36 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 141 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 37 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 21 υπέρ, Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 144 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 38 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 149 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 150 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 26 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 39 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Ε, σχέδιο έκθεση στο σύνολό τη. Να ψηφίσουμε ηλεκτρονικά, παρακαλώ. clearly adopted. Είναι σαφές ότι εγκρίνεται. Mandate, yes. And now we, we are voting the mandate. Uh, Και τώρα ψηφίζουμε για την εντολή. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Επομένως, συγχαρητήρια κύριε Ζαμαρή Καβαντά. Uh, Okay. We uh, continue by... Λοιπόν, συνεχίζουμε με το θέμα 22, ψηφοφορία για την έκθεση ε, του κυρίου Σβιεύκα σχετικά με ε, στάση προς την Κομισιόν για τις διασυνοριακές πτυχές των υιοθεσιών. 118. Τροπολογία 118 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 119 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 8 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 5 6 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 9 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 135 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 136 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 10 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 11 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 11 τόνους μπις υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 5 11 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 12 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 151 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 154 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 155 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 137 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται 126 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 156 υπέρ κατά να ψηφίσουμε ηλεκτρονικά παρακαλώ It has been adopted. Εγκρίνεται. Πέτη 19. Για την πρώτη πρόταση. Υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Για τη δεύτερη πρόταση υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 160. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβιβαστική 13. Υπέρ, κατά αποχές ε, εγκρίνεται 165 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 166 υπέρ κατά αποχές ας ψηφίσουμε ηλεκτρονικά καλύτερα Has been adopted. Εγκρίνεται. 17 bis in favor. 17 bis υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 18 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Ευχαριστώ που ξανάμψατε τα φώτα. 18 υπέρ κατά εδώ θα πρέπει να ψηφίσουμε ηλεκτρονικά. and Απορρίπτεται. 19 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 185 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 20 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 24 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται 200 υπέρ κατά αποχές αποσύρθηκε πάμε συγχωρείτε 201 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 203 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 204 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 205 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 206 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 207 υπέρ κατά. Ας ψηφίσουμε ηλεκτρονικά καλύτερα. Oh, εγκρίνεται. 208 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 209 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Συμβαστική 1 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 4 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται 5 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 6 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 8 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται υπέρ 9 υπέρ συγγνώμη συγγνώμη καταπίπτει 11 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 10, 12, 13 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται συμβιβαστική 2 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 22 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 23 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται συμβαστική 3 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 44 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 4 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 5 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 6 υπέρ κατά εποχές εγκρίνεται 7 υπέρ κατά εποχές εγκρίνεται 48 υπέρ κατά εποχές απορρίπτεται 50 υπέρ κατά εποχές εγκρίνεται 51 υπέρ κατά εποχές εγκρίνεται 54 υπέρ κατά εποχές εγκρίνεται 14 υπέρ συγγνώμη καταπίπτει 57 υπέρ κατά να ελέγξουμε παρακαλώ It is adopted. Εγκρίνεται 58 υπέρ συγγνώμη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 αποχές εγκρίνεται 22 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 94-95 υπέρ κατά να ελέγξουμε παρακαλώ And 96 υπέρ. Κατά. Εποχές. Απορρίπτεται. 97 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 98 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 99 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 100 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 102 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 103-104 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 105 υπέρ κατά να ελέγξουμε παρακαλώ Απορρίπτεται. 6 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 107 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 108 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 110 υπέρ. Κατά. Νομίζω ότι απορρίπτεται, αλλά να ελέγξουμε. Απορρίπτεται. 23 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 116 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 210 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 214 υπέρ. Κατά εποχές εγκρίνεται 213, συγγνώμη καταπίπτει 215 υπέρ κατά εποχές εγκρίνεται 216 υπέρ κατά εποχές απορρίπτεται 217 υπέρ κατά να ελέγξουμε εγκρίνεται 218 υπέρ κατά εποχές απορρίπτεται 219 υπέρ κατά εποχές απορρίπτεται 25 υπέρ κατά εποχές εγκρίνεται 26 υπέρ κατά εποχές εγκρίνεται 27 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 28 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 229 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 230 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 231 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 233 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 237 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 238 υπέρ κατά εποχές απορρίπτεται 2.42 υπέρ κατά εποχές απορρίπτεται 2.41 υπέρ κατά εποχές απορρίπτεται 2.44 υπέρ κατά εποχές εγκρίνεται 2.45 υπέρ κατά πρέπει να το ελέγξουμε Απορρίφθηκε. 2.46 υπέρ. Εποχές απορρίπτεται. 2.47 υπέρ. Κατά. εποχές απορρίπτεται. 2.48 υπέρ. Κατά. εποχές εγκρίνεται. 2.49 υπέρ. Κατά εποχές εγκρίνεται ηλεκτρονικά ψηφίζουμε την έκθεση του συνολό της εγκρίνεται συγχαρητήρια στο κυρίο Βιευκά Now we Τώρα έχουμε την έκθεση του κυρίου Μαστάλκα για την εφαρμογή της οδηγίας του Συμβουλίου 2004 κάθετος 113. Συμβαστική 2 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 11 υπέρ. Κατά. Να ελέγξουμε παρακαλώ. One more vote. Μία ακόμη Εγκρίνεται. Συμβαστική 3. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 15 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 16 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 17 υπέρ. Κατά εποχές εγκρίνεται 19 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται συμβαστική 4 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 23 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 24 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 1 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 2 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται συμβαστική 1 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 5 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 6 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 7 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Ψηφίζουμε το σύνολο της έκθεσης συνολικά, ηλεκτρονικά, με συγχωρείτε. Εγκρίνεται. Συγχαρητήρια στο κύριο Μαστάλκα που δεν μπορούσε να είναι μαζί μας. Τώρα, Έχουμε το σχέδιο γνωμοδότηση για τον έλεγχο τη Μητρώου και τη σύνθεση των ε, ομάδων εμπειρογνωμόνων τη Κομισιόν. Κυρία Κάουφμαν είναι η συγγήτρια. Συμβαστική 1 υπέρ. Κατά αποχέ εγκρίνεται. 4 υπέρ. Κατά αποχέ εγκρίνεται. 5 υπέρ. Κατά. Συγγνώμη. Η 5 καταπίπτει. 6 υπέρ. Κατά αποχές Πρέπει να ελέγξουμε. Εγκρίνεται. Συμβαστική 2 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 3 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 4 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 18 υπέρ κατά εποχές εγκρίνεται 20 υπέρ κατά να ελέγξουμε παρακαλώ εγκρίνεται 5 υπέρ κατά εποχές εγκρίνεται 25 υπέρ κατά εποχές απορρίπτεται 26 υπέρ κατά εποχές απορρίπτεται 27 υπέρ κατά εποχές απορρίπτεται γνωμοδότηση συνολικά ηλεκτρονικά λείπει μία ψήφος Εγκρίνεται. Συγχαρητήρια στην κυρία Κάουφμαν. Και τώρα έχουμε μία ακόμη ενιαία, ψήφο, ενιαία ψηφοφορία ηλεκτρονικά. Άρχεται η ψηφοφορία. Η κυρία που τον έθελε κάτι να πει. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θέλω να διευκρινίσω ότι η σύστασή μου για ψηφοφορία δεν αφορά παρά το σύνολο των κανόνων της αναδιατύπωσης και δεν θα θεωρηθεί ως υποστήριξη στην ουσία αυτής της πρότασης γιατί αντιτίθεμαι κάθετα. Ευχαριστώ. Ας ψηφίσουμε και πάλι ηλεκτρονικά παρακαλώ για το θέμα αυτό. Αναδιατύπωση. Σημείο 27, όπως σας είπα. Σημείο 27. Ακόμη τρεις λείπουν, δεν έχουν ψηφίσει. Λήξη της ψηφοφορίας εγκρίνεται. Συγχαρητήρια στην κυρία Μπουτονέ. Αυτά για τις ψηφοφορίες. Σας ευχαριστώ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 We will continue by the leftovers from... Να συνεχίσουμε με ό,τι μας έχει απομείνει από χτες. Point number 10. Σημείο 10. Και θα ήθελα να δώσω το λόγο στην κυρία Χάνιμπολ να μας κάνει μια αναφορά για την συνάντηση του Διοικητικού Συμβουλίου και της Επιτροπής Προπολογισμών σε σχέση με το Γραφείο Διανοτικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ευχαριστώ. Ήταν ε, μια αξιόλογη συνεδρίαση. Νομίζω ότι είναι πολύ καλό που έχουμε εκπροσώπηση στο Διοικητικό Συμβούλιο, γιατί προφανώς ε, το Γραφείο Διανοητικής Ιδιοκτησίας είναι σημαντικό για μας και να ξέρουμε τι κάνει. Εγώ παρευρέθη εκεί και εκπροσωπούσα την Επιτροπή 15 έως 17 Νοεμβρίου και το Αλικάντε είναι πάντα ευχάριστη τοποθεσία για επίσκεψη. Για να σας αναφέρω ότι συνεδριεκλέξαμε ένα νέο πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και υπήρξε μια ψηφοφορία Συγγνώμη για την προφορά μου στα ισπανικά, μάλλον λάθος το πω το επιθετό της. Την κυρία Πατρίσια Γαρσία Σκουβέρο και εξελέγει γιατί έχει εργαστεί σε όλη της ε, τη ζωή στο Γραφείο Εμπορικών Σημάτων. Έχει σχετική εμπειρία, θεωρώ. Λοιπόν, ότι η συνεδρίαση κυρίως ε, αφορούσε θέματα πρόσληψης προσωπικού και σε αυτή τη συνεδρίαση και στην προηγούμενη συνεδρίαση υπήρξαν κάποια ζητήματα που αφορούσαν την πρόσληψη προσωπικού. Νομίζω ότι βελτιώνονται τώρα. Υπήρχε ένα θέμα για ε, το Συμβούλιο Άσκησης Εφέσεων σε σχέση με το ποιος θα είναι ο πρόεδρος και τώρα θα πάει στο Συμβουλίο για τελική απόφαση, ένα σχέδιο απόφασης για το διορισμό των ε, αρμοδίων αρχών ε, για τον εκτελεστικό διευθυντή. Επίσης, ε, συζητήθηκε αυτό είναι ένα από τα πιο επίμεχα θέματα, όμως βρήκαμε έναν τρόπο να το επιλύσουμε συζητήθηκαν και διάφορες επιλογές για την πρακτική κατανομή μεταξύ των κρατών μελών ε, της αντιστάθμισης του κόστους ε, για τα καθήκοντα που αναλαμβάνουν ε, σε ό,τι αφορά το σύστημα εμπορικών σημάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και υπήρξε και μία κλίδα κατανομής που θα αναφερθεί μετά από τρία χρόνια. Μπορούμε να δούμε λοιπόν πώς θα προχωρήσει αυτό και μια νέα εκδοχή των κατευθυντηρίων γραμμών ε, για τα εμπορικά σήματα παρουσιάστηκαν και συζητήσαμε αυτά στι 15 Νοεμβρίου. Υπήρχε μια κοινή συνεδρίαση τη Επιτροπή Προπολογισμού του Διοικητικού Συμβουλίου 16 και 17 Νοεμβρίου. Στρατηγικό σχεδιασμό για το 2020 παρουσιάστηκε και το σχέδιο εργασία ε, του Γραφείου για το Παρατηρείο υιοθετήθηκε. Συζητήθηκε και υιοθετήθηκε. Αν θέλετε περισσότερε λεπτομέρειε, μπορώ να σα στείλω τα έγγραφα. Η Οργανική Συμφωνία για τη δημοσιονομική πειθαρχία του Δεκεμβρίου 2013 και οι συνέπειε για το γραφείο συζητήθηκαν και ιδίω λόγω των διάφορων θέσεων, των διαφορετικών θέσεων που έχουν το Κοινοβούλιο και η Κομισιόν σε ό,τι αφορά τη χρηματοδότηση και τη στελέχωση των οργανισμών. Νομίζω ότι το ξέρουν τα μέλη της Επιτροπής, όμως ε, δεν ε, μιλάμε μόνο για χρηματοδότηση εδώ, υπάρχει και σημαντικό πλεόνασμα και είναι ένα θέμα συζήτησης. Δεν ξέρω αν ε, η ανησυχία είναι η σωστή λέξη, αλλά πρέπει να γνωρίζουμε ότι η κατάσταση έτσι έχει και μια συμφωνία συνεισφορά στο προπολογισμό ε, του Ευρωπαϊκού Σχολείου στο Λικάντε επιβεβαιώθηκε και θα επαναξεταστεί μετά από τρία έτη. Η, Επιτροπή, η συνάντηση στις 17 Νοεμβρίου της Επιτροπής ε, του Προπολογισμού είχε μια μία έλευση. Δεν ξέρω αν συνάδελφος είναι εδώ και ο κύριος Σεκανόφσκης εξελέγει αντιπρόεδρος της Επιτροπής ε, Προεπιλογισμού ε, από το Φεβρουάριο του 2017 η εφαρμογή του προπλογισμού το 2016 παρουσιάστηκε από το γραφείο και υιοθετήθηκε το πρόγραμμα εργασία για τον προπολογισμό του 2017. στρατηγική κατά της απάτης από το 2017 στο 2020 υιοθετήθηκε και λήφθη μία απόφαση να αγοραστεί ένα αγροτεμάχιο που να ε, συνδέσει τα σημερινά κτίρια με τα κτίρια που είναι υποκατοσκευή προκειμένου να έχουμε ένα ενωπημένο χώρο για τα γραφεία που είναι μάλλον καλή ιδέα γιατί ξέρετε είναι σε πάρα πολύ ωραία τοποθεσία δίπλα στη θάλασσα το κτίριο του γραφείου νομίζω ότι είναι λογικό να επεκταθούν και να επωφεληθούν. Αν έχετε ρωτήσει, ευχαριστώ να απαντήσω. Ευχαριστώ. Θέλει κανένα το λόγο. Όχι. Ευχαριστούμε την κυρία Χάνιμπο για την ε, ενημέρωση αυτή. Ένα άλλο θέμα, το 11 που είχαμε από χτες, είναι μια ενημέρωση για την ερμηνεία και εφαρμογή της διοργανικής συμφωνίας ε, για καλύτερες κανονιστικές ρυθμίσεις. Είμαι συνεισηγητής με τον κύριο Ρίτσαρτ Κομπέτ Θέλω να σε ενημερώσω ότι στις 24 Νοεμβρίου συνεδρίασε για πέμπτη φορά η ομάδα εργασίας. Το κύριο θέμα ήταν η μελέτη αντικτύπου και άλλες δυνατότητες καλύτερης νομοθεσίας. Κάναμε μία ανταλλαγή απόψεων με την Αγγέλικα Νίμπλα και τον Βόλφκαν Χίλα. Όπως ξέρετε, το 2011 η κυρία Νίμπλερ ήταν η συγγήτρια για την ε, εξασφάλιση ανεξαρτήτων ε, μελετών αντικτύπου και ο κύριος Χίμπλερ είναι ο υπεύθυνο για τις μελέτες αντικτύπου και την Ευρωπαϊκή Προστιθέμενη Αξία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ο κύριος Χίλερ μας παρουσίασε τις υπηρεσίε που προσφέρει η διεύθυνσή του που δημιουργήθηκε το 2012 ως συνέχεια της έκθεσης Νίμπλε ο κύριος Χίλερ κυρίως ασχολήθηκε με τις εξάντε μελέτες αντικτύπου η διεύθυνσή του μέχρι στιγμής έχει κάνει γύρω στις 130 ε, αξιολογήσεις των μελετών αντικτύπου και επίκειται και άλλες για μελέτες αντικτύπου που ε, είναι σε φάση εκπόνησης ή μελέτες αντικτύπου που προκαλούν πολλές τροπολογίες από τις κοινοβουλευτικές επιτροπές. Συνήθω γίνονται από εξωτερικές ε, εταιρείες αυτές. Ο κύριος Νίμπλερ είπε ότι οι μελέτες ε, ευρωπαϊκής προσθέμενης αξίας παράγονται από την υπηρεσία του κάθε φορά που το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αρχίζει να συντάσσει εκθέσεις, εκθέσεις πρωτοβουλίας. Μετά από αίτημα της Επιτροπής μας, η διεύθυνσή του άρχισε ένα πιλωτικό πρόγραμμα για να υπάρξει μία πλήρης ε, μελέτη αντικτύπου των εκθέσεων πρωτοβουλίας για το διοικητικό δίκαιο. Επίσης, ο κύριος Χίλερ είπε ότι οι επιτροπές θα έπρεπε να ενθαρρύνονται να καλούν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να υποβάλει τις μελέτες αντικτύπου μαζί με τις αρχικές εξολογήσεις από την υπηρεσία του αυτών των μελετών αντικτύπου. Η κυρία Νίμλερ υπενθύμησε την έκθεση του 2011 ότι πρέπει να είναι ανεξάρτητες αυτές οι μελέτες αντικτύπου και τα αιτήματα που είχε τότε υποβάλει το Κοινοβούλιο. Τόνισε επίσης τη σημασία και των εξάντε αλλά και των εξπός αξιολογήσεων και επένεσε την εργασία της ε, υπηρεσίας του κυρίου Νίμπλερ του κυρίου Χίλερ συγγνώμη θεωρεί όμως ότι οι μελέτες αντικτύπου ναι μεν δεν είναι αρκετά ακόμη αντικειμενικές αλλά γενικά κάνουμε βήματα προς τη σωστή κατεύθυνση. Η κυρία Νίμπλερ χαιρέτησε τα νέα στοιχεία της νέας διοργανικής συμφωνίας για τα θέματα αυτά. Επίσης, θεωρεί ότι το Κοινοβούλιο θα πρέπει να αξιοποιήσει πολύ περισσότερο τις δυνατότητες που έχει για την αξιολόγηση των μελετών αντικτύπου. Όλες οι επιτροπές θα πρέπει να ενθαρρυνθούν να αξιοποιήσουν ε, την υπηρεσία αυτή του Κοινοβουλίου και να χρησιμοποιούν αυτές τις μελέτες αντικτύπου όσο περισσότερο γίνεται. Τόνισε επίσης ότι δεν έχουν γίνει αρκετά από το Συμβούλιο για το θέμα αυτό και ότι το Κοινοβούλιο θα πρέπει να ενθαρρύνει το Συμβούλιο να αξιοποιεί πλήρως τις ε, μελέτες αντικτύπου. Βλέπετε λοιπόν ότι ήταν πολύ χρήσιμη αυτή η συνεδρίαση. Δεν ξέρω θέλει κανείς το λόγο. Δεν βλέπω κανένα. Οπότε, λύγει το θέμα αυτό. Και περνάμε στο σημείο 28 εξέταση σχεδίου γνωμοδότησης για τους κανόνες ασφαλείας και τις προδιαγραφές για τα επιβατικά πλοία. Η εισηγήτριά μας η κυρία Ζωέλ Μπεαζουεγόν. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, πρόκειται για ένα σχέδιο γνωμοδότηση προ την Επιτροπή Μεταφορών και αφορά την ασφάλεια στη θάλασσα για τα επιβατικά πλοία εδώ, στο πλαίσιο του προγράμματο ε, REFIT, η Κομισιόν μα παρουσίασε μια πρόταση οδηγία, παρουσίασε ένα σύνολο προτάσεων, θέτει διάφορε δυνατότητε απλούστευση και εξορθολογισμού του σημερινού ρυθμιστικού πλαισίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης ό,τι αφορά την ε, ασφάλεια των επιβατηγών πλοίων. Ο γενικός στόχος είναι να έχουμε ένα σαφές ε, και επικαιρωμένο και απλό νομικό πλαίσιο των ισχύων των κανόνων, προκειμένου να έχουμε υψηλό επίπεδο ασφάλειας. Ε, διαπιστώνουμε ότι κάποιες διατάξεις που έχουν καθοριστεί από την προηγούμενη οδηγία του 2009 για την ασφάλεια των επιβατηγών πλοίων δεν είναι είναι σήμερα κατάλληλες, δεν χρησιμοποιούνται και επομένως ε, είναι περιτές, είναι συνεκτικές ε, και Παραδείγματο χάρη, δεν φάνηκε απαραίτητο να υποβληθούν ε, τα σκάφη κάτω των 25 μέτρων σε υπονερμένου κανόνε ασφαλεία γιατί είναι υπερβολικά δεσμευτικοί ή δεν μπορούν να εφαρμοστούν. Η καταλληλότητα ορισμένων ορισμών ή διαδικασιών δεν είναι πλέον ε, επίκαιρη και επομένως ε, εδώ συμφωνώ με την Κομισιόν στο σημείο αυτό θα πρέπει να γίνει νέα αξιολόγηση και επικαιροποίηση οι διάφορες ε, στοχευμένες διαδουλεύσεις που έγιναν από την Κομισιόν ε, με εθνικούς εμπειρογνώμονες για την ασφάλεια των επιβατηγών πλοίων καθώς και με ενώσεις ε, επιβατών και με τη βιομηχανία κατέληξαν ότι μία σειρά μέτρων που προτείνονται γίνονται αποδεκτά και θεωρούνται χρήσιμα και εγώ ίδια διαβουλεύτηκα με την Ευρωπαϊκή Ένωση Θαλάσσιας Ασφάλειας, την ΕΜΣΑ, η οποία ουσιαστικά μου είπε τα ίδια. Τώρα, εξέταση της πρότασης οδηγίας που είναι ιδιαίτερα τεχνικού χαρακτήρα. Δεν έχω κάποια αντίρρηση σε αυτό. Ε, και τα σημερινά εδάφια σε ό,τι αφορούν την, την επιτροπολογία είναι σωστά και η διοικητική απλούστευση είναι κάτι που εκτιμάται. Σας προτείνω λοιπόν να εγκρίνουμε την πρόταση χωρίς τροποποίηση. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. Ευχαριστώ πολύ. Ζητά κάποιος το λόγο. Δεν βλέπω κάποιο συνάδελφο να θέλει το λόγο. Ευχαριστώ λοιπόν την κυρία Μπερζέρο. Το επόμενο σημείο είναι η ακρόση για την μεταρρύθμιση του δικαιώματος δημιουργού. Στις 11 έχει προγραμματιστεί. Θα κάνουμε ένα σύντομο διάλειμμα για να μπορούν όλοι να μπουν στην αίθουσα ησύχως και θα ξεκινήσουμε ακριβώς στις 11. Okay, dear colleagues. Συνάδελφοι, νομίζω ότι μπορούμε να ξεκινήσουμε την ακρόαση για τη μεταρρύθμιση των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησία. Σα ευχαριστώ όλους που είστε εδώ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω και τους ε, προσκεκλημένους μας. Σκοπός αυτής της πρώτης ακρόασης είναι να συζητήσουμε την πρόταση οδηγίας για τα πνευματικά δικαιώματα και πιο συγκεκριμένα το ζήτημα του δίκαιου μεριδίου από την αξία. Το άρθρο 13 της προτινόμενης οδηγίας δημιουργεί μια υποχρέωση στους παρόχους ε, διαδικτυακών υπηρεσιών που φιλοξενούν περιεχόμενο που έχουν δημιουργήσει οι χρήστες να χρησιμοποιούν αυτοματοποιημένες τεχνολογίες για τον προσδιορισμό και το φιλτράρισμα των έργων που προστατεύονται από δικαιώματα πνευματική ιδιοκτησίας. Ε, ανακύπτουν διάφορα ερωτήματα. Ποιον αφορά αυτή η υποχρέωση, πώς αυτές οι τεχνολογίες φιλτραρίσματος θα πρέπει να λειτουργούν και είναι αποτελεσματικές. Αυτή η υποχρέωση θα αντιμετωπίσει την το αποκαλούμενο κενό αξίας και θα επαρκεί προκειμένου να εξασφαλίζεται η εφαρμογή των δικαιωμάτων πνευματική ιδιοκτησία. Ποια είναι η σχέση μεταξύ του άρθρου 13 και των διατάξεων ασφαλούς λιμένα της οδηγίας για το ηλεκτρονικό εμπόριο. Για να απαντήσουμε σε αυτά τα ερωτήματα λοιπόν έχουμε προσκαλέσει κάποιου ομιλητέ. Ο πρώτο ε, ομιλητής μας είναι ο κύριο Τομπία Μεκένι, Senior European IP Policy Manager τη Google. Έχετε το λόγο για 10 λεπτά. Καλημέρα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί ε, βουλευτέ, μέλη τη Επιτροπή Νομικών Υποθέσεων. Σα ευχαριστώ για την πρόσκληση που με απευθύνετε. Σήμερα θα ήθελα να δράξω την ευκαιρία για να συζητήσω τρία ζητήματα που νομίζω ότι σχετίζονται με αυτή τη συζήτηση που θα γίνει εδώ σε αυτό το όργανο σε σχέση με το άρθρο 13 συγκεκριμένα. Το πρώτο θέμα είναι πώς η Google ε, καταπολεμά την πειρατεία αλλά ταυτόχρονα δημιουργεί και νέες δυνατότητες ανάπτυξης για τον δημιουργικό τομέα. Πώς εφαρμόζουμε αυτές τις αρχές στις περιπτώσεις, στην περίπτωση μάλλον του YouTube και τρίτον ποιε είναι οι εμπειρίες μας και πώς θα μπορούσαν αυτές να βοηθήσουν ε, το υπόβαθρο και τις, ε, το, γενικότερο πλαίσιο που θα διεξαχθεί τις επόμενες εβδομάδες και μήνες ε, η συζήτηση αυτή εδώ στο Κοινοβούλιο. Η Google λοιπόν καταπολεμά την πειρατεία και βοηθά τους, δικαιούχους, τους κατόχους δικαιωμάτων να παράγουν εισόδημα στο διαδίκτυο. Καταπολεμούμε λοιπόν την πειρατεία ανοιχτά και για τον σκοπό αυτό έχουμε διάφορα μέτρα και πρωτοβουλίες. Έχουμε το Content ID που σχετίζεται και με το YouTube συγκεκριμένα και θα σας το παρουσιάσουμε και στις διαφάνειες. Άλλες διαδικασίες συμπεριλαμβάνουν τις διαδικασίες αφαίρεσης ε, περιεχομένου και την υιοθέτηση στρατηγικών όπως είναι το Follow the Money. Επίσης, δεσμευόμαστε την, ε, στην ε, δημιουργία δυνατοτήτων παραγωγής εισοδήματος για τον δημιουργικό τομέα. Και για να βοηθήσουμε στην καταπολέμηση της ε, πειρατείας, εμείς εφαρμόζουμε μέτρα για την, για την προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας στην Ευρώπη. Το περιεχόμενο λοιπόν μπορεί να προσδιοριστεί και να έχει κανείς πρόσβαση και να το αγοράσει πολλές φορές online, οπουδήποτε σε οποιοδήποτε σημείο στον πλανήτη και σε οποιαδήποτε ε, συσκευή. Έχουμε εταιρικέ σχέσεις με χιλιάδες οργανώσεις, με δισκογραφικές εταιρείε, με ε, εκδότες ε, νέων ε, ειδήσεων, μουσικής, βιβλίων, με μη κυβερνητικές οργανώσεις. Έχουμε λοιπόν δύο βασικές αρχές, την καταπολέμηση της πειρατείας και την μεγέθυνση της αγοράς για τη δημιουργία περιεχομένου στο διαδίκτυο με τρόπο που θα ε, ωφελεί τους ε, κατόχους δικαιωμάτων. Πώς εφαρμόζουμε αυτές τις ε, αρχές, νομίζουμε ότι το κάνουμε με έναν πολύ, πολλά υποσχόμενο τρόπο στο YouTube. Θα ήθελα να σας μιλήσω πρωτού μπω σε λεπτομέρειες τι είναι το YouTube και πώς, ποια είναι η δική μας αντίληψη για αυτή την υπηρεσία. Πρόκειται για μια πλατφόρμα διαμοιρασμού βίντεο, 400 ώρες ε, περιεχομένου ανεβαίνουν κάθε λεπτό. Είναι μια ανοιχτή πλατφόρμα. Καθένας, ο καθένας μπορεί να ανεβάσει βίντεο και να το μοιραστεί με ολόκληρο τον κόσμο μέσω αυτής της πλατφόρμας. Και τρίτον, το YouTube αφορά πολλά περισσότερα πέραν της μουσικής. Είναι πολύ σημαντικό να, κατανοη... να γίνει κατανοητό αυτό, γιατί ε, δεν αφορά μόνο τους παραγωγούς μουσικής το YouTube ο μέσος χρήστης του YouTube θα ακούσει ή θα παρακολουθήσει βίντεο μία ώρα ε, μουσικής τον μήνα. Αυτό ε, ε, ε αν, το, αν το συγκρίνεται με τους ε, πελάτες υπηρεσιών ψηφιακής παροχής μουσικής είναι πολύ πολύ μικρότερο το ποσοστό της μουσικής στο YouTube από ό,τι αλλού. Εδώ ε, εμείς προσπαθούμε δηλαδή να ε, φιλοξενήσουμε διάφορους τομείς του, των δημιουργών στο, στο, στην πλατφόρμα μας ε, κάτι που αφορά εν γέννη τον πολιτισμό και μεταβάλλει και την αντίληψή μας. Υπάρχει για παράδειγμα ε, η, το, η συμφωνική του Βερολίνου που προβάλλει το έργο της μέσω του YouTube και υπάρχουν και νέοι δημιουργοί που έχουν, αποκτούν το κοινό τους μέσω του YouTube ή ο Γεννάτος Προτζούρ που ε, βάζει στο, ανεβάζει στο YouTube ντοκιμαντέρ για την γη ε, ή και άλλες ε, οργανώσεις οι οποίες προωθούν και προβάλλουν το έργο τους μέσα, μέσω του YouTube της πλατφόρμας μας. Λοιπόν, να σας δώσω κάποια Πώς ε, λοιπόν ε, εφαρμόζουμε αυτές τις ε, αρχές, τις δύο αρχές, πολέμηση πειρατείας και δημιουργία ευκαιριών για τους δημιουργούς. Ε, πέραν του YouTube Red, το οποίο είναι μια συνδρομητική υπηρεσία του YouTube, ε, ο βασικότερος τρόπος ε, δημιουργίας εισοδήματος στο YouTube αφορά την ε, κατοχήρωση δικαιωμάτων και εισοδήματος μέσω διαφημίσεων στο YouTube που κατευθύνονται στους δημιουργούς. Τρία δισεκατομμύρια δολάρια έδωσε στους δημιουργούς τον τελευταίο χρόνο η YouTube στους δημιουργούς. Χρησιμοποιούμε λοιπόν τις διαφημίσεις. Ε, ε, πώς μπορεί κανείς όμως να παράγει εισόδημα με το δικό του κανάλι ή με περιεχόμενο που έχει δημιουργήσει ο χρήστης. Είναι, είναι διαφορετικά πράγματα. Το, ίδιο, το, το κανάλι που ανήκει σε κάποιον ε, ανήκει στον ίδιο το χρήστη. Εκεί μπορεί να αποφασίσει αν θέλει να ε, ενεργοποιήσει τις διαφημίσεις ή όχι και μέσω αυτού του τρόπου μετά λαμβάνει το μεγαλύτερο μέρος των διαφημιστικών εσόδων. Αυτή είναι η μία. Ε, ε, εκδοχή. Η άλλη εκδοχή είναι το περιεχόμενο των, που δημιουργείται από τους ε, χρήστες. Εκεί θα μιλήσουμε και το Content ID. Εκεί, εδώ έχουμε να κάνουμε την περίπτωση όπου ο χρήστης ανεβάζει βίντεο στο YouTube που περιλαμβάνει και περιεχόμενο που ανήκει σε κάποιον άλλων. Σε αυτές τις περιπτώσεις ε, δίνουμε τη δυνατότητα στους δημιουργούς να επιτρέψουν την παραμονή αυτού του υλικού στην πλατφόρμα και να αποκτήσουν εισόδημα μέσω αυτού του περιεχομένου που έχει δημιουργηθεί από άλλους χρήστες. Ε, πριν από ε, κάποια χρόνια μπορούσε κανείς να πει ότι το περιεχόμενο που δημιουργούνταν από χρήστες ήταν μια μορφή ε, πειρατείας. Γι' αυτό και εμείς δημιουργήσαμε το Content ID για την καταπολέμηση πειρατείας στο διαδίκτυο. Το Content ID λοιπόν προσδιορίζει, ταυτοποιεί ε, περιεχόμενο που προστατεύεται από πνευματική ιδιοκτησία και δίνει τη δυνατότητα στο δημιουργό του να τον μπλοκάρει σε περίπτωση που θέλει. 98% των, ε, της διαχείρισης πνευματικών δικαιωμάτων στο YouTube πραγματοποιείται μέσω του Content ID ε, είναι ένα εργαλείο που πραγματικά με πολύ γρήγορο και αποτελεσματικό τρόπο διαχειρίζεται το περιεχόμενο που είναι πάρα πολύ μεγάλο ε, αλλά μας δίνει και τη δυνατότητα να ανταποκρινόμαστε στις νομικές μας υποχρεώσεις, να ελέγχουμε το περιεχόμενο που ανεβαίνει στην πλατφόρμα μας. Φυσικά το YouTube ε, και το Content ID είναι περισσότερα από μια απλή εφαρμογή ε, εκτέλεσης και κατοχύρωσης δικαιωμάτων. Πολλοί δημιουργοί επιλέγουν να μην μπλοκάρουν πλήρως το πλήρως το δικό τους υλικό σε βίντεο άλλων, αλλά επιλέγουν την, ε, την δυνατότητα να επιτρέψουν τα βίντεο αυτά να συνεχίσουν να εμφανίζονται στην πλατφόρμα μας και να λαμβάνουν ένα εισόδημα από, τις από τα διαφημιστικά έσοδα. Ε, θα μπορούσε λοιπόν αυτό που παλιότερα μπορούσε να θεωρείται πειρατεία πλέον φαίνεται ότι είναι οικονομική δυνατότητα γιατί είναι ένας πολύ πρακτικός τρόπος να παράγει κανείς εισόδημα για τον εαυτό του με βάση το δικό του υλικό και μέσω του περιεχόμενου που δημιουργεί άλλος. Ε, έτσι λοιπόν απλουστεύονται και οι διαδικασίες γιατί για παράδειγμα το μισό του εισοδήματος που παράγεται στο YouTube προέρχεται από ε, περιεχόμενο που παράγουν οι ίδιοι οι χρήστες, ακόμη και για τις δισκογραφικές εταιρείες. Λοιπόν, πώς λειτουργεί το Content ID, γιατί νομίζουμε ότι μπορούμε να αντλήσουμε κάποια σημαντικά διδάγματα, μας έχει διδάξει, εν πάση περιπτώσει, κάποια, πράγματα όσον αφορά την εφαρμογή τέτοιου λύσεων. Εδώ, λοιπόν, ε, ξαναλέω, ε, είναι απόλυτα σαφή τα πράγματα. Ο κατόχος ενός δικαιώματος των δικαιωμάτων μπορεί να μπλοκάρει ε, ένα ανέβασμα ή μπορεί να αποτιμήσει αυτό το περιεχόμενο του βίντεο που έχει χρησιμοποιήσει, που έχει δημιουργήσει άλλος για να το, σε, χρήματα, για να το αποτιμήσει σε, χρήματα για τον εαυτό του. Εδώ βλέπετε την ροή εργασιών, στα, δεξιά βλέπετε το, το ε, ένα βίντεο για παράδειγμα που χρησιμοποιεί ένας ε, φαν ε, εδώ μπορεί το Content ID το εντοπίζει και δίνει τη δυνατότητα στον κάτοχο των δικαιωμάτων αν θέλει να τον μπλοκάρει ή να το αφήσει στην πλατφόρμα. Έτσι λοιπόν λαμβάνει ένα ε, αρχείο ο κάτοχος του δικαιώματος ε, με, ε, όπου μάλιστα μπορεί και να κάνει διάφορες επιλογές για το πού μπορεί να προβάλλεται, με ποιον τρόπο κτλ. Ε, οι επιλογές ε, ε, που, που δίνονται είναι σαφείς και δεν επιδέχονται καμία αμφισβήτηση. Τέλος θα ήθελα να αναφερθώ και σε κάποιες προκλήσεις που έχουμε αντιμετωπίσει κατά την εφαρμογή του Content ID στο YouTube. Ε, σας είπα ότι είναι κάτι πάρα πολύ θετικό γιατί ε, οι φαν από πειρατέ έχουν γίνει μια πηγή εσόδων για την μουσική βιομηχανία ε, μας επιτρέπει την δυνατότητα ε, να διαχειριζόμαστε το πολύ περίπλοκο ζήτημα της ποικιλία που υπάρχει στην ε, μουσική βιομηχανία. Το Content ID βεβαίως έχει προσαρμοστεί και με βάση τις εξελίξεις, ε, εντοπίζει soundtrack, βίντεο και μουσικές συνθέσεις. Αυτό σημαίνει ότι σήμερα όταν για παράδειγμα μπορεί να τραγουδάτε ένα τραγούδι και το βάζετε αυτό στο YouTube η μελωδία μπορεί πραγματικά να εντοπιστεί και να ενημερωθεί ο κάτοχος των δικαιωμάτων αυτού του τραγουδιού. Υπάρχει λοιπόν ένας ανταγωνισμός σε αυτόν τον, ε, ε, τεχνολογιών. Ε, υπάρχουν βέβαια και οι χρήστες οι οποίοι προσπαθούν να αποφύγουν ή να ε, κοροϊδέψουν κατά κάποιον τρόπο τα, τις τεχνολογίες αυτές. μπορεί κανείς, ε, όπως στην, σε μια εικόνα μπορείς να αλλάξεις για παράδειγμα τον κορεσμό, ε, έτσι προσπαθούν διάφοροι χρήστες να παραλλάξουν λίγο το περιεχόμενό τους προκειμένου να διαφεύγουν από τα δίχτυα και τα φίλτρα του Content ID. Πάντως αυτό που έχει σημασία είναι να ε, εντοπίζεται πάντοτε η σωστή ισορροπία ανάμεσα στα δικαιώματα των κατόχων των δικαιωμάτων και των χρηστών της πλατφόρμας. Γιατί αυτό που θέλουμε να επιτύχουμε είναι το YouTube να παραμείνει ε, ανοιχτή πλατφόρμα ε, δίνοντας ε, στους δημιουργούς τη δυνατότητα να προστατεύουν τα δικαιώματά τους. Γι' αυτό το σκοπό χρειάζεται και κίνητρα, χρειάζονται και κίνητρα προκειμένου να εξασφαλίζονται αυτές οι αρχές. Σε 30 δευτερόλεπτα τελειώνω κύριε Πρόεδρε αν, αν μου τα παραχωρείτε. Λοιπόν, πρώτον, τεχνολογία δεν μπορεί να εντοπίσει αν δικαίως ένας κάτοχος δικαιωμάτων ε, προσφεύγει ε, κατά ενός χρήστη. Έχει συμβεί, για παράδειγμα, ε, στο παρελθόν να έχουν συμβεί τέτοιες περιπτώσεις. Επίσης, η τεχνολογία δεν θα πρέπει να είναι υποχρεωτική γιατί πρέπει να υπάρχει δυνατότητα και στους χρήστες να προσφεύγουν κατά ε, αξιώσεων αφαίρεσης από, το, από την πλατφόρμα μας. Βρίσκεται σε, σε εξέλιξη βέβαια η όλη διαδικασία, είναι, μεταβάλλεται διαρκώς αυτή η, ε, αυτή η τεχνολογία, γι' αυτό και εμείς δεν θα θέλαμε να... Ε, στηρίξουμε μια γενική καθολική εφαρμογή μιας τέτοιας λύσης ε, σε όλο τον ε, κλάδο. Ευχαριστώ πολύ. Δεύτερος ομιλητής είναι ο κύριος Τιρί Σεβιάρ, Γενικός Διευθυντής της Blue Efficiency. Δέκα λεπτά. Έχετε το λόγο. Bonjour. Καλημέρα σας. Σας ευχαριστώ που μας καλέσατε να παρουσιάσουμε τις δραστηριότητές μας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και θα σας ε, δώσω κάποιες αποσαφηνήσει για την καταπολέμηση της πειρατεία ε, και από τη σκοπιά του νόμου και από τη σκοπιά της ε, δικής μου εταιρείας. Η Blue είναι μια εταιρεία που ιδρύθηκε το 2008 είναι μια γαλλική startup τεχνολογίας ε, η οποία ε, ήθελε να προστατεύσει τα ε, άτομα στην καθημερινή τους μάχη κατά της πειρατείας. Εμείς προστατεύουμε και τους κατόχους δικαιωμάτων και τα έργα τους και εργαζόμαστε αποκλειστικά στο τομέα του οπτικοακουστικού με οριζόντιο τρόπο. Δηλαδή, προστατεύουμε τα έργα τους ε, ε, όταν εμφανιστούν στο ίντερνετ και καθ' όλη τη διάρκεια ζωής τους στο διαδίκτυο και λαμβάνουμε κάθε απαραίτητη πράξη έρευνα εντοπισμού των παραβάσεων και απόσυρσης των έργων. Ε, απλώς χρειάζεται να μας δώσουν μια εντολή και κατόπιν εμείς κάνουμε μια διαδικασία προστασίας επί, της πλατφόρμας. Είναι συνεχής ο ρόλος μας και φυσικά ο στόχος είναι να έχουμε την ε, συντομότερη απόσυρση ε, των ε, έργων και να καταστούν όσο δυνατόν πιο σπάνια. Μιλάμε για έργα που παράνομα έχουν μπει στο διαδίκτυο. Οι δράση μας βασίζονται σε δύο πυλώνες. Καταρχήν στη τεχνολογία, θα την αναπτύσσουμε στον οίκο μας και είναι καρπός της έρευνας και της ανάπτυξής μας και έχει ως στόχο να υπάρχει συνεχής πλοήγηση στο ίντερνετ και εις βάθος προκειμένου να εντοπίσουμε όλες τις παραβάσεις ε, δικαιωμάτων δημιουργού ε, για τους πελάτες μας. Ο δεύτερος πυλώνας είναι η περάσπιση του νόμου ανάλογα με την επικράτεια όπου γίνονται οι παραβάσεις. Εμείς βασιζόμαστε στο δίκαιο, φυσικά στο ευρωπαϊκό δίκαιο και στην Αμερικανική DCMA, η οποία παρακολουθείται σε παγκόσμιο επίπεδο, τηρείται σε παγκόσμιο επίπεδο και στις Ηνωμένε Πολιτείε ε, οι περισσότεροι από τους ε, οποίους, στους οποίους απευθυνόμαστε ζητούν την εφαρμογή της Αμερικανικής νομοθεσίας. Οι πελάτες μας ε, είναι ακόμη και τηλεοπτικά κανάλια, συγγραφείς, εκδότες ε, έχουμε το χάρη τη UGC Images, ε, ε, διεθνεί εταιρείε ή εταιρείε όπω που μας ζητούν μελέτες και επίσης έχουμε και την Ακαδημία Σέζαρ και επίσης ε, έχουμε και πελάτες όπως πολύ γνωστά φεστιβάλ στον κόσμο του κινηματογράφου και μέσα και μέλη της ΦΙΚΑΜ της ε, Ομοσπονδίας Βιομηχανιών του Κινηματογράφου στην Γαλλία έχει ισχυρό ρόλο και ε, ουσιαστικά εφαρμόζει το γαλλικό δίκαιο τώρα για την προστασία σύμφωνα με την Blue Efficiency εδώ θα συμφωνήσω με όσοι υπόθηκαν από τον εκπρόσωπο της Google. Έχουμε την ε, χρήση των αποτυπωμάτων. Εμείς υλοποιούμε αποτυπώματα για να προστατεύσουμε καλύτερα ε, τα έργα στο YouTube ε, και αλλού. Πρόκειται για αποτυπώματα που γίνονται για το Content ID ή με την υπογραφή INA. Υπάρχει και το Audible Magic στις Ηνωμένε Πολιτείε και δημιουργούμε και διαχειριζόμαστε αυτά τα αποτυπώματα. Είναι μια δουλειά καθημερινή και παραδείγματο χάρη δεν, έχουν, δεν υπάρχουν πάντα οι αρμοδιότητες για να αντιμετωπιστούν τα θέματα της επικράτειας και της σύγκρουσης μεταξύ επικρατιών. Τώρα, βλέπουμε πότε εμφανίζεται μια πειρατική πηγή στο διαδίκτυο και τότε αναλαμβάνουμε την εργασία προστασίας και ε, εργαζόμαστε στις πλατφόρμες όπου ε, έχουμε περιεχόμενο που δημιουργείται από το χρήστη και περιλαμβάνουμε τα βίντεο ε, που προσπαθούν ουσιαστικά να ξεπεράσουν τα φίλτρα και θέλουμε τελικά να αποσύρουμε αυτά τα βίντεο. Σε ό,τι αφορά τώρα τις ιστοσελίδες αναφοράς, ε, όπου είναι αφιερωμένες ε, στην ε, πειρατεία, εκεί αυτές οι ιστοσελίδες είναι αυτές που δημοσιεύουν κάποιους συνδέσμους φιλοξενίας, δηλαδή μιλάμε για πλατφόρμες φιλοξενίας, έχουμε περίπου 100 και ουσιαστικά πρόκειται για πειρατεία σε δύο επίπεδα, δηλαδή δεν υπάρχει ευρετηρίαση ε, και στο περιεχόμενο ε, ουσιαστικά δεν υπάρχει ευρετηρίαση. Επίσης, ε, αποσύρουμε κάποιες ευρετηριάσεις των ε, μηχανών αναζήτησης που οδηγούν προς ε, τα έργα και εδώ Έχουμε κάποια κοινωνικά δίκτυα που μπορούν να συνδέουν σε περιοδικές ιστοσελίδες, αλλά ε, σιγά σιγά διάφορα τέτοια μέσα κοινωνική δικτύωση, όπως στο Facebook επιτρέπουν στους χρήστες να διαθέσουν ολόκληρο το περιεχόμενο. Το δεύτερο στάδιο είναι ουσιαστικά να χαρακτηρίσουμε τις, ε, παρεμβα... τις παραβάσεις. Ε, αυτό γίνεται είτε αυτόματα είτε χειρονακτικά. Έχουμε διάφορα τεχνικά μέτρα που μπορούμε να προτείνουμε. και το τρίτο στάδιο είναι οι διαδικασίες απόσυρσης που μπορεί να γίνουν μέσω διεπαφών ε, όπως πρότεινα το YouTube είτε μέσω ψηφιακών ε, κοινοποιήσεων. Ουσιαστικά εδώ μιλάμε για μια πολύ γρήγορη απόσυρση ή μπορεί ε, ουσιαστικά να βάλουμε ένα δικηγόρο ε, να παρέμβει αν έχουμε ουσιαστικά υποτροπή στην παράβαση. Έχω σημειώσει κάποια στοιχεία κλειδιά για την πειρατεία, αλλά πολύ γρήγορα θα περάσω στις αντιδράσεις μου απέναντι στην οδηγία. Καταρχήν, η πειρατεία αφορά όλα τα είδη των έργων, των οπτικοακουστικών, είτε παλιά είτε καινούρια, κάθε είδους, όπως σας είπα. Εμείς εκτιμούμε ότι έχουμε περίπου 100 πλατφόρμες φιλοξενίας όπως είναι το YouTube αλλά και κάποιες άλλες πλατφόρμες που μαζικά ε, προβαίνουν σε διάθεση έργων παράνομα και κάθε εβδομάδα ανοίγει μια καινούργια ιστοσελίδα για την ευρετηρίαση αυτών των ιστοσελίδων φιλοξενίας και καθημερινά βλέπουμε ε, χιλιάδες ουσιαστικά διαθέσεις κάθε έργο και ένας στους δέκα δεν προβαίνει στην απόσυρση. Έτσι λοιπόν εδώ μιλάμε για ανθρώπους που έχουν συνείδηση ε, για το τι κάνουν και η προθεσμία απόσυρσης γίνεται είτε αμέσως αλλά μπορεί να πάρει και αρκετές μέρες. Εδώ. Θέλω να σας πω ποια είναι η γνώμη μου απέναντι στην οδηγία και κυρίως ε, τι συμβαίνει ακριβώς με τον κόσμο της πειρατείας ε, σήμερα. Οι πλατφόρμες ε, ουσιαστικά όπως το YouTube είναι η κορφή του παγόβουνου. Οι τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται είναι πάρα πολύ αποτελεσματικές, δεν υπάρχει αμφιβολία και Πρέπει να συμφωνήσω με το YouTube όταν λέει ότι όταν υπάρχουν πειρατικά βίντεο που διαπερνούν τα φίλτρα πρέπει να γίνει, γίνεται μάλλον μια πραγματική δουλειά για τη βελτίωση των τεχνικών. Όμως πάντοτε έχουμε βίντεο που συχνά λιώνονται και μπορούν ε, να διαπεράσουν τα φίλτρα. Ε, γίνεται ε, ουσιαστικά κάποια αλλίωση των χαρακτηριστικών. το χάρη μπορεί να γίνεται επιτάχυνση στις σκηνές του βίντεο και εγώ σας μιλούσα πριν το χάρη για το μέρος του παγώνου που βρίσκεται κάτω από το νερό. Έχουμε, το χάρη, κάποιες πλατφόρμες οι οποίες δεν κάνουν ευρετηρίαση του περιεχομένου. Και εδώ έχουμε την ουσία του προβλήματος, την ουσία της πειρατείας. Δεν είμαι πεπισμένος ε, ότι στοχεύονται αυτές από την ε, οδηγία ε, που έχει σχεδιαστεί. μέτρα φιλτραρίσματος όπως έχουν ε, προταθεί στην οδηγία που δεν γίνονται από ανάλυση του περιεχομένου όπως το Content ID είναι πάρα πολύ ισχυρά και μπορεί να έχουν σημαντικό αντίκτυπο. Όμως, αν ε, αφήσουμε ελεύθερες τις πλατφόρμες να θεσπίσουν τα μέτρα που επιθυμούν, θα μπορούσαν να υιοθετήσουν ένα μέτρο φίλτρου που να αφορά το περιεχόμενο, αλλά αυτό θα αφήσει να περάσουν πάρα πολλά πράγματα. Υπάρχουν στο διαδίκτυο αρκετοί αλγόριθμοι για την ανάλυση του περιεχομένου και αυτό είναι ο κίνδυνο σε σχέση με την εισαγωγή μέτρων φιλτραρίσματος. Και για να ολοκληρώσω, τα μέτρα που κατά την άποψή μας και την εμπειρία μας θα ήταν πιο απλά ε, είναι ε, ουσιαστικά κάποια στάδια με, για την αναγνώριση του περιεχομένου που για μας είναι κάτι πολύ ισχυρό. Υπάρχει κάτι πολύ απλό οι πλατφόρμες φιλοξενίας μπορούν να δράσουν γρήγορα για την απόσυρση του περιεχομένου και θα πρέπει να υπάρχουν πρόσθετες υποχρεώσεις σε σχέση με την ταχύτητα, δηλαδή κάτι πιο συγκεκριμένο, γιατί κάποιες αποσύρουν το ίδιο λεπτό και μπορούν να αποσύρουν το ίδιο λεπτό, δεν ε, υπάρχει λοιπόν λόγος να μην μπορούν να το αποσύρουν και ολοκληρώνω σε 30 δευτερόλεπτα η διάθεση φίλτρων με απλή υπογραφή. Δηλαδή δεν χρειάζεται απαραίτητα να έχουμε υπογραφές με αναγνώριση περιεχομένου, αλλά απλές υπογραφές αρχείων που δεν έχουν εφαρμοστεί ποτέ, αλλά μπορεί να έχουν ισχυρό αντίκτυπο στην καταπολέμηση της πειρατείας. Αυτό θα ήταν ε, ένα πραγματικό στάδιο καταπολέμησης. Δεν βρίσκω τη λέξη, λέει ο μιλτής αλλά θα μπορούσαν ε, αυτά ουσιαστικά να συμπεριληφθούν μέσα σε μια οδηγία. Πάντως και η αναγνώριση του περιεχομένου επί της ουσίας είναι μια αποτελεσματική διαδικασία. Σας ευχαριστώ. Thank you very much. Ευχαριστώ πολύ. Ακούσαμε λοιπόν την άποψη των παρόχων ε, υπηρεσιών διαδικτύου και των startup. Μπορούμε να τις συζητήσουμε αυτές τις δύο παρουσιάσεις αν οι συνάδελφοι θα ήθελαν ε, να κάνουν ερωτήσεις, να σχολιάσουν τις δύο πρώτες παρουσιάσεις που ακούσαμε. Υπάρχει να δυνατότητα. Η κυρία Κομοντίνε. Ευχαριστώ. Έχω κάποιες ερωτήσεις δύο μάλλον ερωτήσεις για την Google και τις άλλες δύο για το Blue Efficiency. Πρώτη ερώτηση. Αν σας πούν να αφαιρέσετε περιεχόμενο, παραμένει μονίμως εκτός. Τι γίνεται, γιατί μία από τις ανησυχίες και τα, τις διαμαρτυρίες που ακούμε είναι όταν αναφερείτε περιεχόμενο, γιατί σας το λέει το Content ID, την επόμενη μέρα κάποιος άλλος το ξανανεβάζει. Και πρέπει να επαναληφθεί η διαδικασία. Έτσι έχουν τα πράγματα. Ή ο μηχανισμός αυτός Content ID μαθαίνει πλέον να αναγνωρίζει αυτό το περιεχόμενο και αμέσως να το ξανααφαιρεί εάν ξανανεύει. Δεύτερη ερώτηση που αφορά και τους δύο μάλλον ε, ομιλητές μας. Λέμε για την ε, διανομή του εισοδήματο μεταξύ των ε, επιγραμμικών πλατφορμών και των ε, κατόχων δικαιωμάτων. Αλλά θεωρώ ότι μπορεί να ενδιαφέρονται για το κέρδος, την αξία που παίρνουν, που παίρνουν το περιεχόμενό τους από τη χρήση του. Θα έπρεπε λοιπόν η πρόταση της Επιτροπής να κάνει μια προσπάθεια να ε, αυξηθεί η διαφάνεια στην αλυσίδα αξίας. Υπάρχει ενδεχόμενα ε, κοινή χρήση στοιχείων, όπως για παράδειγμα αναλυτικών στοιχείων, που θα μπορούσαμε να δώσουμε στους ε, κατόχους δικαιωμάτων για να δούμε πώς θα διαμορφώσουμε τις διατάξεις περί διαφάνειας. Είπατε ότι ο μηχανισμός Content ID δεν αναγνωρίζει αν ο χρήστης έχει χρησιμοποιήσει σωστά το περιεχόμενο το οποίο προστατεύεται από πλευρά πνευματικών δικαιωμάτων με βάση και τις εξαιρέσεις. Απαντούν οι κάτοχοι δικαιωμάτων λέγοντας ναι, ναι, μπορεί να παραμείνει γιατί υπάρχουν εξαιρέσεις. Και με βάση εξαιρέσεις μπορώ εγώ ως χρήστης να το χρησιμοποιήσω αυτό το περιεχόμενο. Και η Google λέει ότι χρειάζονται 6 ώρες για να επεξεργαστούν ένα αίτημα για αφαίρεση περιεχομένου. Αλλά η Blue Efficiency είπε ότι καμιά φορά χρειάζονται και δύο μέρες μέχρι να αφαιρεθεί το περιεχόμενο. Γιατί υπάρχει αυτή η διαφορά. Μπορείτε να μας εξηγήσετε. Ευχαριστώ. Η κυρία Ρέντα. Ευχαριστώ πολύ για τις παρουσιάσεις σας. Ο στόχος μας είναι η νομοθεσία να είναι σαφής, να μπορεί να εφαρμοστεί εύκολα. Στον κύριο Σεβιλιά, καταρχάς. Είπατε ότι εφαρμόζεται τον Ευρωπαϊκό Νόμο για τα, για τα διανοτικά δικαιώματα. Εφόσον στέλνετε ειδοποιήσεις για αφαίρεση περιεχομένου, λαμβάνετε υπόψη τις εξαιρέσεις στα διανοτικά δικαιώματα ποιων χωρών εάν κάποιο κάτοχο δικαιωμάτων είναι στη Γαλλία, αλλά ο χρήστη που έχει ανεβάσει περιεχόμενο είναι στη Γερμανία και η πλατφόρμα ε, εδρεύει ε, ε, στην Ιρλανδία. Ποιες εξαιρέσεις ισχύουν. Στέλνετε ένα, μια ειδοποίηση για τα διανοητικά δικαιώματα και περιμένετε η πλατφόρμα να εφαρμόσει τις διατάξεις. Κύριε Μακένι, είπε τα προβλήματα που έχουν αυτές οι αυτόματες, ε, ε, τα αυτόματα λογισμικά αναγνώρισης του, των διανοητικών δικαιωμάτων και τι περιορισμούς έχουν. Κάποιες ειδοποιήσεις που εστάλησαν οδήγησαν ε, στην αφαίρεση περιεχομένου και τελικά διαπιστώθηκε ότι το 17% του περιεχομένου που κατέβηκε, που αφαιρέθηκε, έγινε λανθασμένα. Πώς μπορεί να βελτιωθεί. Μήπως αυξηθεί το πρόβλημα με την επέκταση της χρήσης αυτών των αυτοματοποιημένων λογισμικών. Και επίσης, η πρόταση της Επιτροπής λένε ότι οι πάροχοι πλατφορμών πρέπει να ενημερώνουν τους κατόχους για τα ποσοστά επιτυχίας της τεχνολογίας τους. Έχετε στοιχεία για αυτά τα ποσοστά πόσο συχνά η τεχνολογία σας αναγνώρισης περιεχομένου δεν αναγνωρίζει το περιεχόμενο. Η κυρία Νίμπλα. Ευχαριστώ. Μια σύντομη παρατήρηση και μια ερώτηση και στους δύο ομιλητές μας. Ευχαριστώ για τις ε, παρουσιάσεις σας. Παρατήρηση. Η πρόταση της Επιτροπής για τα δυνατικά δικαιώματα λέει ότι η παραγωγή, η δημιουργή, οι κάτοχοι πρέπει να ενισχυθούν και να κερδίζουν και αυτοί από αυτή τη διαδικασία. Ε, συμφωνείτε ότι αυτός είναι ο στόχος της πρότασης της Κομισιόν, ότι θα οδηγήσει σε αυτό το αποτέλεσμα. Μιλήσατε για πειρατεία και οι δύο. Παλιότερες, ε, παλιότερου και, ναι, και πρόσφατου περιεχομένου ποιο είναι, ποιος είναι ο όγκος της πειρατείας που διαπιστώσατε. Είναι περιφερειακά φαινόμενα ή η πειρατεία είναι όντως πρόβλημα. Ε, Mrs. Η κυρία Γκέριγκερ. Ευχαριστώ πολύ για τις παρουσιάσεις σας. Να ρωτήσω κάτι που σχετίζεται και με αυτά που μόλις ακούσαμε από την κυρία Νίμπλα. Ποια είναι η οικονομική διάσταση της πειρατείας. Ε, αυτές που μπορέσατε να εντοπίσετε. Και πόσο ε, σημαντικά είναι τα πρόστιμα. ύψους για περιπτώσεις παραβίασης ε, δικαιωμάτων. Καταλαβαίνω ότι υπάρχει εδώ θέμα και εμπορικού απορρίτου. Αλλά θα ήθελα να έχω μια ιδέα για την τάξη μεγέθους. Θέλουμε ο κανονισμός. Θέλουμε η νομοθεσία που θα εγκρίνουμε να προλαμβάνει τέτοια φαινόμενα στο μέλλον. Θέλουμε να δούμε λοιπόν ποιες είναι οι τάξεις μεγέθους ε, οικονομικές και τι προσδοκίες υπάρχουν επίσης. Αυτών που θέλουν να αντιμετωπίσουν την πειρατεία. Οι προσδοκίες αυτών που θέλουν να γίνει γνωστό, να δημοσιευθεί το περιεχόμενό τους. Έχουμε κολλήσει μια αφίσα που λέει θα υπάρξει μεταρρύθμιση αλλά για μένα είναι μικρή σημασία, διακοσμητικές αυτές οι, οι αλλαγές. Ποιες είναι οι ουσιώδεις ε, προσδοκίε που έχουμε. Σας παρακαλώ να δώσετε σύντομες ερωτήσει. γιατί δεν έχουμε χρόνο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και ευχαριστώ και για τις ερωτήσεις. Πρώτα να ξεκινήσω με το ερώτημα της, του, του καταμερισμού των εσόδων και των κερδών. Πρώτον, να πω ότι πιστεύουμε ότι το YouTube είναι ένας καθαρός ε, συμβάλλον ε, όσον αφορά τα έσοδα από τον δημιουργικό τομέα. Όσον αφορά την τον διαμορισμό των κερδών εμείς θέλουμε να ε, διευρύνουμε αυτόν τον διαμερισμό μέσω του ψηφιακού περιεχομένου ε, και είναι πολύ ενδιαφέρον ότι αυτό ήδη συμβαίνει γιατί πολλές από τις υπηρεσίες μας ε, ε, όπως το YouTube ε, επιστρέφει τον, το μεγαλύτερο μέρος των διαφημιστικών εσόδων του, από, προς τους δημιουργούς. Άρα ε, όσο περισσότερα χρήματα βγάζει το YouTube, τόσο περισσότερα χρήματα βγάζουν οι δημιουργοί, τόσο περισσότερα χρήματα βγάζουμε και εμείς. Ε, σας είπα ότι 3 δισεκατομμύρια ήταν ε, τα έσοδα για τη μουσική βιομηχανία, 2, 2 δισεκατομμύρια για το περιεχόμενο από χρήστες. Αυτό βέβαια δεν είναι στατικό, ε, αντιθέτως ε, θέλουμε να διευρύνουμε αυτά τα ποσά. Αν δείτε το παρελθόν, στο YouTube υπάρχει μια πολύ σαφή και σταθερή τάση των επιστροφών των διαφημιστικών δαπανών που επιστρέφονται στους δημιουργούς 50% και πάνω. Ε, επίσης συμμετέχουμε σε άλλες ε, πρωτοβουλίες όπως είναι το YouTube Red, μια συνδρομητική επιπληρωμή υπηρεσία που έχει ξεκινήσει τη λειτουργία της στις ΕΠΑ προς το παρόν. Αυτό που, ε, το θέμα που τέθηκε σε σχέση με τα δεδομένα είναι πάρα πολύ σημαντικό και ανοίγει μια περαιτέρω συζήτηση για το πώς θα μπορούσε να βελτιωθεί αυτή η, η αξία. Το YouTube έχει εργαλεία για να ε, μοιράζεται δεδομένα με τους εταίρους, δηλαδή του, ε, δηλαδή το, άτομο που κατέχει ε, τα δικαιώματα πνευματικής δικαιοσύνης ενός υλικού, έχει πρόσβαση στο ποιο, ποιο υλικό του, από ποιον και σε τι συχνότητα έχει ε, ε, χρησιμοποιηθεί. Το Content ID δίνει μια τέτοια δυνατότητα για παράδειγμα, να μην υπάρχουν διαφημίσεις, αλλά να συλλέγονται αυτά τα δεδομένα και μόνο. Θα μπορούσα να σας δώσω και ένα παράδειγμα. Αν έχετε ε, μια ευρωπαϊκή ταινία, για παράδειγμα, θα υπάρχουν άνθρωποι στην Νότια Αμερική που παρακολουθούν αυτό το υλικό σας. Θα μπορούσε κανείς λοιπόν να ζητήσει δικαιώματα ε, χρήσης ε, σε, για αυτούς τους ανθρώπους. Ε, θα μπορούσε ίσως ε, με αυτόν τον τρόπο να δημιουργηθούν διάφορες πηγές εισόδου και στις Φιλιππίνες ακόμη. Υπάρχουν, υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη συζήτηση για το πώς θα μπορούσε να λειτουργήσει εύρυθμα και ομαλά η ογαρά, αλλά ο όρος γι' αυτό είναι να υπάρχουν ίση όροι και ίση πρόσβαση στα δεδομένα. Προς το παρόν έχουμε δυνατότητα ε, παροχής αυτών των πληροφοριών μόνο στους ε, εταίρους μας, αλλά υπάρχει ένα ευρύτερο ζήτημα για το πώς μπορούν να ρέουν αυτές, αυτά τα δεδομένα σε όλη την ε, έκταση της αλυσίδας αξίας, κάτι που επιδιώκεται και με αυτή την πρόταση, η οποία επίση ενισχύει την διαφάνεια. Αυτά ως προς τον διαμορισμό των κερδών και της αξία είναι ένα από τα ζητήματα που είναι πάρα πολύ σημαντικά. Για το δεύτερο θέμα, που αφορά τη χρήση περιεχομένου και των ε, τεχνολογιών ε, διαχείρισης του περιεχομένου όπως το Content ID. Το Content ID δεν αφορά μόνο το μπλοκάρισμα αλλά αφορά και την δημιουργία νέων ευκαιριών για τους ε, κατόχους και τους χρήστες να δημιουργήσουν νέες, νέο εισόδημα. Δύο είναι οι αντιλήψεις. Πρέπει να ομολογήσουμε ότι η τεχνολογία δεν μπορεί να αναγνωρίσει τις εξαιρέσεις ε, στα δικαιώματα πνευματικής ε, ιδιοκτησίας. Γι' αυτό και εμείς σκεφτόμαστε πώς μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε, τι είδους εχέγγυα μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε στο πλαίσιο αυτών των τεχνολογιών, γιατί αυτή τη στιγμή δεν γίνεται. Δεν υπάρχει δυνατότητα να ενταχθεί μια τέτοια λειτουργία στο, στο λογισμικό αυτό. Στοιχεία. Τα, οι αξιώσεις του Content ID ε, μπορούν να τύχουν τις προσφυγής των ε, χρηστών, δηλαδή οι χρήστες μπορούν να προσφύγουν ε, κατά των αποφάσεων του που λαμβάνει αυτό το Content ID και οι περιπτώσει αυτές ανέρχονται στο 1%. Αυτό σημαίνει για τη μουσική βιομηχανία ότι μιλούμε για περίπου 2.000-3.000 ε, χρήστες που προσφεύγουν κατά αξιώσεων Content ID. Δεν είναι λοιπόν αμελητέ αυτές, αυτοί οι αριθμοί. Οι χρήστες φαίνεται ότι ε, ενδιαφέρονται πολύ για το υλικό του και ε, βεβαίως αντιδρούν όταν θεωρούν ότι μία ε, αξίωση είναι άδικη ή αθεμελίωτη. Ε, φυσικά εδώ πρέπει να σκεφτούμε πώς, που, που μπορούν να, να, σε ποια κατεύθυνση θα κινηθούν οι διαφημιστικές δαπάνες. Ε, πάντως αυτό που μας ενδιαφέρει είναι ότι ένας χρήστης που λαμβάνει αξίωση να μπορεί να προσφύγει κατά αυτής. Ο χρόνος εξαρτάται ε, από διάφορους παράγοντες. Ε, όταν δεν υπάρχει συμφωνία χρήστη και κατόχου δικαιωμάτων, τότε ο κάτοχος δικαιωμάτων οφείλει να υποβάλει επίσημο αίτημα ε, αφαίρεσης και μάλιστα θα προσφύγει δικαστικά εναντίον του χρήστη για τη χρήση του υλικού του. Ε, επίσης, ε, εμείς έχουμε χρηματοδοτήσει τις περιπτώσεις ορισμένων χρηστών οι οποίοι θέλουν να ε, καταπολεμήσουν δικαστικά αξιώσεις που έχουν υποβληθεί εναντίον τους. Όσον αφορά την πειρατεία, θα ήθελα να επαναλάβω και να τονίσω ότι εμείς ε, αντιμετωπίζουμε το θέμα αυτό ανοιχτά. Θέλουμε να είμαστε αποτελεσματικοί αλλά και αναλογικοί. Εμείς επεξεργαζόμαστε εκατομμύρια αιτήματα με πάρα πολύ υψηλε ταχύτητες μέσω του Content ID που ε, υπερβαίνει και τις απαιτήσει της νομοθεσίας προκειμένου όλοι οι κάτοχοι δικαιωμάτων να έχουν τα απαραίτητα μέσα στα, στη διάθεσή τους προκειμένου να διαχειρίζονται τα δικαιώματά τους και τον τρόπο που χρησιμοποιούνται στο ίντερνετ. Ευχαριστώ. Σε ό,τι αφορά την εκχρημάτιση των ε, έργων, οι κάτοχοι δικαιωμάτων ε, στο 90% δεν ε, εκκληματίζουν τα έργα τους στο διαδίκτυο. Βρίσκονται δηλαδή σε μια διαδικασία ε, η παραγωγή τηλεοπτικών σειρών ή ταινιών βρίσκονται σε μια διαδικασία μη εκκληματισμού. Τώρα δεν θα είχα απάντηση να σας δώσω αλλά να κάνω ένα σχόλιο όταν ε, ένα βίντεο σε μια πλατφόρμα όπως ε, το YouTube περνά μέσα από ε, μια ταινία γιατί έχει αλλάξει η μορφή του, έχει αλλοιωθεί η μορφή του για άλλους λόγους, κάτι που είναι ανήθικο αλλά συμβαίνει και θα αναφερθώ και στον όγκο εδώ της πειρατείας, μπορεί πολύ εύκολα να φτάσει σε δεκάδες, εκατοντάδες χιλιάδες θεάσεις και μερικές φορές δεν είναι σπάνιο να δούμε ένα βίντεο που θα ξεπεράσει το εκατομμύριο θεατές. Και αυτό οφείλεται στο ότι κάποιος ε, πειρατής έχει θέσει το περιεχόμενο επιγραμμικά και έχει βάλει και διαφήμιση. Και αυτό που κάνουν οι κάτοχοι των δικαιωμάτων ε, λένε ναι το έχουμε αποσύρει αλλά όλα τα έσοδα από τη διαφήμιση που πέρασε τελικά από τα διάφορα φίλτρα, αυτά τα έσοδα από τη διαφήμιση γιατί δεν έρχονται σε μένα και πού πηγαίνουν. Μία παρατήρηση λοιπόν που λαμβάνουμε είναι αυτή πολύ συχνά και δεν έχω συγκεκριμένη απάντηση. Τώρα για τα άλλα ζητήματα για το θέμα της προθεσμίας, είπα ότι χρειάζονται σε κάποιες περιπτώσεις περισσότερες μέρες και σε κάποιες πλατφόρμες του YouTube η απόσυρση ε, για ένα βίντεο που έχει περάσει από φίλτρα μπορεί να γίνει ή επειδή δεν υπάρχει αποτύπωμα που να έχει ε, υλοποιηθεί από εμά, αυτή η απόσυρση γίνεται άμεσα. Δεν ε, υπάρχει καμία εμφιβολία, κάνουμε μια άμεση δράση. Τώρα, σε ό,τι αφορά τις προθεσμίες ε, της απόσυρσης, ε, αυτό έχει να κάνει με τον κύριο όγκο του προβλήματος, δηλαδή με τις εκατοντάδες πλατφόρμες φιλοξενίας ε, που δεν προβαίνουν σε ευρετηρίαση και μαζικά ε, ουσιαστικά καταγράφονται και χρησιμοποιούνται από τους πειρατές ε, για να διαθέσουν το περιεχόμενο ορισμένοι ε, θα αποσύρουν αμέσως αλλά ορισμένοι θα πάρουν και το χρόνο τους. Όπως σας είπα, ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να χρειαστούν τρία λεπτά, σε άλλες περιπτώσεις τρεις μέρες. Αυτό είναι ένα πραγματικό πρόβλημα. Και αυτό έχει να κάνει με την μαζική πτυχή της πειρατείας σήμερα. Είναι η προβληματική της δραστηριότητας της πειρατείας. Ε, τώρα, να απαντήσω για τον όγκο. Ανέφερα κάποιους όγκους, μπορεί να υπάρχουν στο YouTube, όμως ε, σε ό,τι αφορά τον κύριο όγκο του προβλήματος, ε, δηλαδή όχι την κορφή του παγόβουνου, όταν κάνουμε κάποιες μελέτες παρακολούθησης ε, φτάνουμε σε ταινίες ή σε δεκάδες, εκατοντάδες ε, χιλιάδες θεάσεις ε, ή λήψεις αρχείων. Είναι δύσκολο να αναλύσουμε και να προβάλλουμε όλα αυτά τα στοιχεία, τα ελάχιστα αριθμητικά στοιχεία σας αναφέρουμε εδώ, είναι μαζικός ο χαρακτήρας και όλα τα περιεχόμενα γίνονται αντικείμενο πειρατείας ανάλογα με την εμπορική τους επιτυχία. Και οι μελέτες που μπορέσαμε να κάνουμε με ένα άτομο που ε, ουσιαστικά ζητούσε βίντεο video demand ε, τελικά ε, είχαν κάνει μια παράνομη κατανάλωση και αυτό εξηγεί τι γίνεται στην αγορά των βίντεο, σε ό,τι αφορά την εξαίρεση από τα δικαιώματα δημιουργού. Σε πλατφόρμες όπως το YouTube ή άλλες πλατφόρμες, τα συστήματα, με τα συστήματα που υπάρχουν, γίνεται, υπάρχει δυνατότητα να διαχειριστεί κανείς ε, τις ε, εδαφικές εξαιρέσεις και επιτρέπει στους χρήστες του ίντερνετ ε, που έχουν δει ένα βίντεο ε, να το αποσύρουν ε, ή μπορεί να δουν ένα τμήμα παραδείγματος χάρη μιας εκπομπής. Έχουμε τη χρήση την εφαρμογή του Fair και στην περίπτωση αυτή που έχουμε το Fair δεν αποσύρεται το βίντεο. Εμείς λέμε ότι είναι γενικά αποδεκτό το Fair και οι τεχνικές που τίθενται σε εφαρμογή για να ε, ε, αντιμετωπίσουμε τα αιτήματα γενικά γίνονται αποδεκτές. Σας είπα ότι έχουμε εκατοντάδες πλατφόρμες φιλοξενίας που κατά 50-80% χρησιμοποιούνται μοναδικά, ε, συγγνώμη, χρησιμοποιούνται μόνο για να διατεθούν εκεί παράνομα περιεχόμενα αν ε, κάποια στιγμή του στείλουμε μία κοινοποίηση, πρόκειται ε, ουσιαστικά για ολόκληρε ταινίε ή για ολόκληρε ε, σειρέ, και οι, κάτοχοι των δικαιωμάτων δεν θέλουν σε καμία περίπτωση να τα δουν όλα αυτά στο διαδίκτυο και τελικά ποτέ δεν λαμβάνουμε μία απάντηση, γιατί απέναντί μα έχουμε πειρατές, απλού πειρατέ. Και ουσιαστικά, όπως σας είπα, θα πρέπει να δούμε και τα δύο τμήματα ε, και ε, την κορφή του παγόμενου που έχουμε παράνομο περιεχόμενο, αλλά ε, και ό,τι βρίσκεται ουσιαστικά στον κύριο όγκο του προβλήματος, τα μαζικά τα παράνομα περιεχόμενα. Ευχαριστώ. Τώρα περνάμε στο δεύτερο μέρος της ακροασής μας, να ακούσουμε την άποψη των κατόχων δικαιωμάτων, των χρηστών, των δημιουργών. Έχουμε τρει ομιλητέ. Σας παρακαλώ να μην μιλήσετε πάνω από 8 λεπτά για να μας μείνει κάποιος χρόνο για συζήτηση γιατί αλλιώ δεν θα μας μείνει. Ο κύριος Αγκουστίν Ρέινα από την οργάνωση BUC είναι η Ευρωπαϊκή Οργάνωση Καταναλωτών. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ και τη Γραμματεία για την πρόσκληση. Θα επιχειρήσω να είμαι πολύ σύντομο. Η οργάνωσή μα εξετάζει τα, τα διανοητικά δικαιώματα από δύο πλευρές. Πρώτα απ' όλα η διαθεσιμότητα και η πρόσβαση ε, των καταναλωτών σε νόμιμες προσφορές και από την άλλη μεριά οι παραβιάσεις. Έτσι προσπαθούμε να εξετάσουμε το θέμα. Δεν θα σας πω κατά πόσο υπάρχει το λεγόμενο κενό αξίας ή όχι. Αυτό είναι η εμπορική πλευρά. Οι συνάδελφοι ξέρουν περισσότερα από μένα. Εγώ θα μιλήσω για την επίπτωση της πρότασης Επιτροπής του άρθρο 13 στους καταναλωτές. Υπάρχουν τρία βασικά προβλήματα με την προσέγγιση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το κενό αξία. Πρώτα απ' όλα, ασυμβατότητα με το ενωσιακό δίκαιο, ιδιαίτερα με την οδηγία για το ηλεκτρονικό εμπόριο. Δεύτερον, ανεπαρκή ε, εγγυήσει για τους καναλωτές και τρίτον ενδεχόμενες παραβιάσεις της νοσιακής χάρτας ε, θεμελιωδών δικαιωμάτων. Πρώτα απ' όλα, συμβατότητα με τον νοσιακό νόμο. Πρώτα απ' όλα, να εξετάσουμε το πρώτο άρθρο της πρώτης οδηγίας, όπου επίτρες δεν περιλαμβάνεται η οδηγία για το ηλεκτρονικό εμπόριο ως ένα από τα μέσα που δεν επηρεάζεται από αυτή την οδηγία. Αυτό είναι πολύ σημαντικό γιατί δείχνουν ότι υπάρχει σαφής πρόθεση να επηρεαστεί ο τρόπος εφαρμογής αυτής της οδηγίας, ιδιαίτερα μέσω του άρθρου 13 της νέας οδηγίας. Αυτό το άρθρο 13 επιβάλλει υποχρέωση να εγκριθούν τεχνολογίες αναγνώρισης περιεχομένου που σύμφωνα με την ε, νομολογία του δικαστηρίου θα μπορούσαν να θεωρηθούν ως υποχρέωση επιτήρηση σε σχέση με το άρθρο 15 της οδηγίας για το ηλεκτρονικό εμπόριο. Πρέπει να ε, λάβουμε υπόψη ότι αυτή η διάταξη εγκρίθηκε για να αναπτυχθεί το διαδίκτυο με στόχο να βοηθήσει την ανάπτυξή του. Αν συνδυάσουμε αυτή την υποχρέωση με την παράγραφο 2 της αιτιολογικής σκέψης 38, μπορούμε να θεωρήσουμε ότι υπάρχει ένα νέο καθεστώς ευθύνης και για την οδηγία ηλεκτρονικού εμπορίου. Γιατί στην ουσία είναι ερμηνευτικός κανόνας που θα υπεδείκνει στο δικαστή πότε ένας πάροχος υπηρεσιών μπορεί να αξιοποιήσει τις εξαιρέσεις από την ευθύνη του άρθρου 14. Αυτή η αιτιολογική σκέψη 38 αντανακλά την ε, νομολογία στην ε, απόφαση ε, L'Oreal eBay, παράγραφος 116. Εάν ένας πάροχος βελτιώνει ή κάνει διαφήμιση για κάποιο έργο, ανεξάρτητα από τη φύση, μπορεί να έχει επιπτώσεις στο πώς αξιολογούμε τον ενεργό ρόλο της πλατφόρμας. Δεν θα μπορούσε να αξιοποιήσει δηλαδή την εξαίρεση από την ε, ευθύνη. Αυτό αποκλίνει και από την ομολογία, όπως είπα, σε συγκεκριμένη περίπτωση, αλλά και από την οδηγία για το ηλεκτρονικό εμπόριο, που λέει ότι ο πάροχος, για να μην μπορεί να ωφεληθεί από τις εξαιρεσει, πρέπει να γνωρίζουν το περιεχόμενο. Γιατί αυτό έχει έννοια για του καταναλωτές. Αν οποιαδήποτε πλατφόρμα είναι υπεύθυνη για το περιεχόμενο που ανεβάζουν οι καταναλωτές, αυτό σημαίνει περαιτέρω περιορισμοί. Το βλέπουμε ήδη στην απόφαση Δέλφη εναντίον Εστονία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Αυτό θα δημιουργήσει νομική ασάφεια. Δεν θα ξέρω ποιο είναι υπεύθυνο γιατί. Γιατί αυτό θα εξαρτάται απόλυτα από την ερμηνεία ενό δικαστή για το πώ ερμηνεύει το, την αιτιολογική σκέψη 38 σε σχέση με τι διατάξει τη ε, οδηγίας για το ηλεκτρονικό εμπόριο. Και αυτό θα μπορούσε να επιβάλλει και άλλες υποχρεώσεις επιτήρησης άλλων παρόχων. Και αυτός ήταν ο κύριος στόχος ε, της ε, ε, επιβολής σεβασμού ανθρωπίνων δικαιωμάτων και δεν θέλω να κοινολογώ, αλλά θεωρώ ότι θα σταματήσει να υπάρχει το ίντερνετ όπως το ξέρουμε. Αν θα πρέπει οι ιδιωτικοί φορείς να ελέγχουν το περιεχόμενο που περνάει από τους παρόχους ηλεκτρονικών υπηρεσιών. Τώρα για το άρθρο 13 λέγεται ότι τα κράτη-μέλη θα δημιουργήσουν μηχανισμούς προσφυγής και ε, παραπώνων εάν δεν συμφωνούν με την ε, λειτουργία αυτών των τεχνολογιών από πλευράς καταναλωτών θεωρούμε ότι υπάρχει άλλο πρόβλημα. Πρώτα απ' όλα είναι λύση ex post, γιατί το περιεχόμενο έχει ήδη αφαιρεθεί θα είναι πολύ δύσκολο να εφαρμοστεί γιατί στα διανοτικά δικαιώματα δεν έχουμε δικαιώματα των χρηστών αλλά εξαιρέσεις. Πώς λοιπόν αυτές οι νέες τεχνολογίες θα λάβουν υπόψη τις εξαιρέσεις και μόλις τώρα μάθαμε ότι τα λογισμικά που ήδη λειτουργούν δεν μπορούν να το επιτελέσουν αυτό. Ως δικηγόρος για θέματα καταναλωτών οι μηχανισμοί προσφυγής δημιουργούνται για να ασκηθεί ένα δικαίωμα. Αλλά η εξαίρεση είναι άλλου τύπου. Είναι πολύ δύσκολο να προβλέψουμε πώς θα λειτουργήσει στην πράξη αυτό. Τι θα γίνει για παράδειγμα εάν κάτι δεν καλύπτεται από μια εξαίρεση. Τα κράτη, συγγνώμη, τα μέλη μας σε 10 διαφορετικές χώρες κάναμε μια ε, έρευνα Μιλήσαμε με υπουργεία, με ειδήμονες για τέτοια θέματα για να μάθουμε πώς ε, αντιμετωπίζουν αυτή την πρακτική των καταναλωτών. Είναι νόμο ένας καταναλωτής, για παράδειγμα, ένας για παράδειγμα να μοιραστεί σε μια κοινωνική πλατφόρμα ένα αεραστεχνικό βίντεο από πίσω ακούγεται μια, ένα τραγούδι. Και η απαντήση ήταν σαφής αλλά μετά αφήνουμε την ε, αξιολόγηση του, της νομιμότητας στις ε, τεχνολογίες αυτές και σε ένα μηχανισμό προσφυγής που δεν ξέρουμε πώς θα εφαρμοστεί στην πράξη. Τρίτο σημείο. Παραβίαση των ε, θεμελιωδών δικαιωμάτων, ενδεχόμενα. Σύμφωνα με μια περίπτωση Σαμπάμ vs. Netlog, η διατάξεις του άρθρου 13 είναι ασύμβατες με τρία δικαιώματα. Ελευθερία της επιχειρηματικότητας, ελευθερία στην προστασία των προσωπικών δεδομένων και η ελευθερία έκφρασης και ενημέρωσης. Αυτό που μας εκπλήσει είναι ότι στην μελέτη επιπτώσεων η Επιτροπή αναγνωρίζει ότι μπορεί να έχει επίπτωση αυτή η νέα οδηγία στην ελευθερία έκφρασης και ενημέρωσης. Αλλά αυτό που είναι ιδιαίτερα αξιοσημείωτο, θεωρούν ότι αυτή η αρνητική επίπτωση απαλύνεται από τις εγγυήσει που προτείνουν και άλλες που ήδη λειτουργούν. Βλέπουμε λοιπόν ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή οι αρνητικές επιπτώσεις σε σχέση με την άσκηση των θεμελιωδών δικαιωμάτων είναι κάτι το οποίο νομικά δεν μπορεί να εφαρμοστεί και ταυτόχρονα η χρήση αλγορίθμων στις διάφορες πλατφόρμες δεν λαμβάνουν υπόψη τα θεμητά, τις θεμητές μορφές χρήσης από πλευράς των καταναλωτών και σύν της άλλης έχουν αποδειχθεί ήδη ανεπαρκή. Ο προηγούμενος συνάδελφος είπε ότι το 1% είναι το ποσοστό το οποίο είναι υπό αμφισβήτηση. Αλλά αν δείτε πραγματικά το πεδίο στο οποίο ασκείται αυτό. Αυτό σημαίνει ότι στο 1 ένα εκατομμύριο οι 10.000 έχουν προβλήματα σε σχέση με τη λειτουργία του συστήματος. Εγώ σαν δικηγόρος, αν δω ότι ένα τέτοιο ποσοστό, ένα τέτοιο αριθμός πελατών δεν είναι ικανοποιημένος, αυτό σημαίνει ότι το σύστημα είναι σαφές ότι είναι ανεπαρκές. Λοιπόν, η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε επίπεδο νομικό είναι αμφισβητήσιμη. Οι ρήτρες προστασίας των καταναλωτών είναι ανεπαρκέστατες. Το άρθρο 13 είναι σαφώς εναντίον της νομολογίας του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου και υπάρχει μια επίγουσα έκκληση να εξεταστεί εκ νέου η πρόταση αυτή σε σχέση με την Χάρτα των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων. Κάτι θα πρέπει να γίνει λοιπόν και θα πρέπει να βρούμε λιγότερο παρεμβατικές λύσεις όπως οι εθελοντικές συμφωνίες και οι κατευθυντήριες γραμμές για την σωστή εφαρμογή του άρθρου 14. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. από την Ένωση των Ανεξαρτήτων Εταιριών Παραγωγής Μουσικής. Παρακαλώ να σεβαστείτε το χρόνο που έχετε στη διάθεσή σας. Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Αντιπροσωπεύουμε περίπου 4.000 μικρομεσαίες επιχειρήσεις στην Ευρώπη. 80% των επενδύσεων και των θέσεων εργασίας. Θα ήθελα να σας δώσω την δική μας προοπτική για την συγκεκριμένη πρόταση. Um, today we have και σε σχέση με το λεγόμενο value gap, τις διαφορές δηλαδή στην καθαρή αξία. Υπάρχει ένα πρόβλημα με τον τρόπο λοιπόν τον οποίο δημιουργείται αυτό το value gap. Η δυτική μουσική στην παρούσα φάση δεν μεταφράζεται σωστά σε σχέση με το μέγεθός της σε επίπεδο αξίας και γι' αυτό πολλές φορές ο τρόπος με τον οποίο κατεβάζει κανείς μουσικής καταστρέφει την δημιουργία και καταστρέφει επίσης και στρεβλώνει τον ανταγωνισμό και σε σχέση με άλλες επίσημες πλατφόρμες κατεβάσματος μουσικής. Υπάρχουν ποσοστά λοιπόν τα οποία μονομερώς καθορίζονται από τις πλατφόρμες φόρτωσης, είτε δέχεται κανείς ο εκπρόσωπος των παραγωγών αυτά τα επίπεδα αποζημιώσεων, είτε δεν θα κυκλοφορήσει από, τα συγκεκριμένες, από τις συγκεκριμένες πλατφόρμες η μουσική του. Δεν είναι σωστή λειτουργία της ελεύθερης αγοράς και δεν μπορεί κανένας να βγάλει την αξία των προϊόντων του όπως θα έπρεπε. Για να καταλάβετε λοιπόν την το μέγεθος του προβλήματος μετά από έρευνες της IPI το 2015 υπήρξαν 900 εκατομμύρια άνθρωποι που άκουσαν και κατέβασαν μουσική με έσοδα 634 εκατομμυρίων, κάτι το οποίο θα πρέπει να συγκριθεί στις υπηρεσίες συνδρομής όπου μόνο 68 εκατομμύρια απέδωσαν 2 δις και αυτό θα πρέπει να συγκριθεί και με τον αριθμό που έδωσε το bias. Αυτό είναι ένα ποσό το οποίο εκπροσωπεί ουσιαστικά και το YouTube από μόνο του σε σχέση με την παραγωγή μουσικής τα τελευταία 10 χρόνια. Δηλαδή ε, τρεις φορές ε, το κανονικό έσοδο από το κατέβασμα μουσικής ε, μέσω των συγκεκριμένων συνδρομών. Οι άνθρωποι που χρησιμοποιούν το YouTube σήμερα σαν βασικό, βασική πηγή μουσικής. Δεν ψάχνουν να βρουν νέα μουσική, στην ουσία κατεβάζουν τη μουσική την οποία γνωρίζουν. Και αυτό δημιουργεί προβλήματα στη νέα παραγωγή. Τι θέλουν τα μέλη μας. Καταρχάς θέλουν τα μέλη τους να πληρώνονται σωστά. Είναι κάτι το οποίο είναι προς όφελος των μελών μας και των καλλιτεχνών γενικότερα να διατίθεται η μουσική τους με την, στην ευρύτερη δυνατή εμβέλεια. Θέλουν να διαπραγματεύονται τα ποσοστά της χρήσης της μουσικής τους και θέλουν φυσικά αυτοί που θέλουν τη μουσική τους να μπορούν να τα κατεβάζουν. Σήμερα το 80% των εσόδων των μελών από τις πλατφόρμες αυτές προέρχονται από τα έσοδα τα οποία πληρώνουν ουσιαστικά οι χρήστες δεν θέλουν ε, να αυξηθεί το κόστος, θέλουν ένα μεγαλύτερο ποσοστό από τα έσοδα. Το σύστημα αυτό λοιπόν πρέπει ε, με σωστές διαπραγματεύσεις να αμύψει σωστά τους παραγωγούς. Πιστεύουμε ότι η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι ένα καλό πρώτο βήμα έτσι ώστε να διευκρινιστεί η κατάσταση στην αγορά ιδιαίτερα σε σχέση με τις μεγάλες πλατφόρμες. Νομίζω ότι έχουμε μια ξεκάθαρη δυνατότητα να τεθεί τέλος στα προβλήματα της αγοράς ή σε κάποια από αυτά και να μπορέσουν οι ε, παραγωγοί να εισπράξουν τα σωστά έσοδα από τα προϊόντα τους. Πώς θα γίνει αυτό. Ε, καταρχάς διευκρινίζεται <clears throat> το τρόπος λειτουργίας των υπηρεσιών κατεβάσματος μουσικής μέσω συμφωνιών, κάτι που θα επιτρέψει στους παραγωγούς και δημιουργούς και κατόχους δικαιωμάτων να λειτουργήσουν σε καλύτερο επίπεδο. Υπάρχει, υπηρεσία για υπάρχει υποχρέωση για τις υπηρεσίες αυτές να πάρουν τα κατάλληλα μέτρα προστασίας με τη σωστή τεχνολογία των έργων τα οποία διαθέτουν. Τώρα σε σχέση με την δακτυλοσκόπηση, εμείς έχουμε, επαναλαμβάνω, την υποχρέωση να παρακολουθούμε ε, τον τρόπο με τον οποίο γίνονται ε, αυτές οι διαδικασίες κατεβάσματος μουσικής. Νομίζω ότι έτσι και αλλιώ μπορούμε να βασιστούμε στις βάσεις δεδομένων οι οποίες γνωστοποιούνται και με τις οποίες ενημερώνονται οι κάτοχοι δικαιωμάτων. Και δεν χρειάζονται νέα μέσα όπως ε, το obligation Νέες μέθοδοι, εν περιπτώσει, παρακολούθησης των διαδικασιών κατεβάσματος. Διαδικασίες παρακολούθησης λοιπόν αυτών οι οποίοι κατεβάζουν τη μουσική δεν θα πρέπει να ξεπεράσουν ένα κάποιο επίπεδο περιπλοκότητας. Θα πρέπει λοιπόν οι διαπραγματεύσεις να ξεκινήσουν κάτι το οποίο θα καταστήσει ικανά τα μέλη μας να διαπραγματεύονται σωστά με τις πλατφόρμες. Ε, θα πρέπει επίσης έτσι να αποτρέψουμε και το στρεβλό ανταγωνισμό ανάμεσα σε κάποιες από τις υπηρεσίες οι οποίες λειτουργούν ε, ε, ελλειπτικά σε επίπεδο νομικό και υπηρεσίες πλατφόρμες όπως το Spotify το οποίο λειτουργεί με βάση συμφωνίες με τις ενός παραγωγών. Έτσι θα γνωρίζουν και οι καταναλωτές ότι οι αγαπημένοι τους παραγωγοί πληρώνονται σωστά όταν χρησιμοποιούνται οι υπηρεσίες τους και τα προϊόντα τους. Θα πρέπει να δημιουργήσουμε λοιπόν ένα μη στρεβλό περιβάλλον. Thank you very much. Ευχαριστώ πολύ. Τελευταίος ομιλητής είναι η κυρία Σιλβή Φοντόρ από το Κέντρο για τη Βιομηχανία Εικόνας. Έχετε το λόγο. Οκτώ λεπτά, αν μπορείτε, σας παρακαλώ. Ευχαριστώ. Λοιπόν, εκπροσωπώ την βιομηχανία εικόνας και φωτογραφίας, μια, ένα από τα θύματα της ε, διαδικτυακής πειρατείας, όπως θα δείτε. Η παρουσίασή μου αφορά πρώτον το value gap για τον ε, κλάδο μας και συνέχεια θα μιλήσω για την οδηγία. Όσον αφορά αυτό το, τη διαφορά αξίας, ε, εμείς ε, στον κλάδο μας πολλές φορές το αποκαλούμε και value block, γιατί οι κάτοχοι των δικαιωμάτων δεν λαμβάνουν κανένα εισόδημα. Υπάρχει λοιπόν μια ε, διαφορά μεταξύ ζήτησης και εσόδων. Κάποια στοιχεία να σας δώσω. Στο πλαίσιο αυτής της οδηγίας, το 85% των εικόνων που εμφανίζονται ε, στο διαδίκτυο αποτελούν παράνομες, παράνομα αντίγραφα. Αυτό αφορά το άρθρο 13, όπου ε, αντίστοιχες διατάξεις ε, βρίσκονταν σε ισχύ 10-15 ε, χρόνια και ήταν πολύ αποτελεσματικές, αλλά το, το κόστος ε, το επομίζονται μόνο οι κάτοχοι των δικαιωμάτων. Είναι ένα επιχειρηματικό μοντέλο στην ουσία το οποίο ε, ε, σπάει στην ουσία την αλυσίδα αξίας. Είναι ένα μοντέλο το οποίο χρησιμοποιείται από τις πλατφόρμες προκειμένου να προσελκύσει χρήστες, τους προσελκύει, χρησιμοποιεί δεδομένα αυτών των χρηστών για να έχει διαφημιστικά έσοδα. Και από αυτά τα διαφημιστικά έσοδα ούτε ένα σεντ δεν πηγαίνει προς τους κατόχους των δικαιωμάτων. Εδώ βλέπετε τα διάφορα social media. Εδώ μπορείτε να δείτε μια ε, παράνομη χρήση μιας εικόνας ενός βατράχου στο Pinterest, ε, εδώ λεοπαρδάλης, ε, ό,τι θέλετε. Παντού βρίσκονται εικόνες όπου συλλέγονται στις πλατφόρμες αυτές τεράστιες ποσότητες εικόνων και φωτογραφιών δίνουν τη δυνατότητα του διαμοιρασμού και της κοινή χρήση. Αλλά αυτό δεν είναι πρόβλημα. Αλλά το πρόβλημα είναι ότι τα τελευταία χρόνια δημιουργούνται και λειτουργίες προκειμένου να παραμένουν οι χρήστες στο... στη δική τους ιστοσελίδα και να μην παραπέμπονται στην ε, αρχική ε, ιστοσελίδα από την οποία έχουν προέλθει οι φωτογραφίες. Εδώ βλέπετε ε, την εξέλιξη του Google Images. Πάνω βλέπετε την παλιά εκδοχή η οποία ακόμη βρίσκεται σε ισχύ και σε λειτουργία στη Γαλλία και κάτω βλέπετε την βελγική εκδοχή του Google Images. Παρόμοια είναι τα πράγματα και σε άλλες χώρες όπως τη Γερμανία. Βλέπετε ποια είναι η διαφορά. Ε, πάνω η εικόνα ε, εμφανίζεται μεγάλη και ταυτόχρονα εμφανίζεται στο παρασκήνιο και η ιστοσελίδα από την οποία έχει προέλθει ε, η εικόνα αυτή. Ενώ στη δεύτερη, στο, ε, στο δεύτερο στιγμιότοπο βλέπετε ότι όλες αυτές τις πληροφορίες έχουν αφαιρεθεί χωρίς να υπάρχει τίποτα στο παρασκήνιο. Με αυτόν τον τρόπο η Google ε, κατάφερε να διατηρεί τους χρήστες ε, στη δική της πλατφόρμα. Πάνω κάτω μπορεί κανείς να σκρολάρει και να δει παρόμοιες εικόνες. Άρα οι χρήστες δεν αναγκάζονται να φύγουν από το Google γιατί καδράρονται οι εικόνες που έχουν αναζητήσει εντός του Google. Και έτσι δεν καταλήγουν ποτέ στους πραγματικούς κατόχους, στις ιστοσελίδες των πραγματικών κατόχων, των δικαιωμάτων αυτών των φωτογραφιών. Γενικά, Όσον αφορά την οδηγία, θεωρούμε ότι είναι ένα καλό πρώτο βήμα, γιατί αποκαθιστά ε, ίσους όρους ε, για όλους τους εμπλεκόμενους φορείς. Με τον, ε, ε, ενθαρρύνει την συνεργασία και δίνει κίνητρα στη χρήση τις τεχνολογίες. Εμείς δεν ε, υποστηρίζουμε την υποχρεωτική χρήση τέτοιου είδους τεχνολογιών. Εμείς θέλουμε να δοθούν κίνητρα, γιατί αυτή τη στιγμή δεν έχουμε καμία σχέση με τις ε, εκάστοτε πλατφόρμες και ούτε ενδιαφέρονται εκείνες να έρθουν σε συνεργασία μαζί μας. Όσον αφορά την ε, τεχνολογία, θα ήθελα και εγώ να θέσω ένα ερώτημα στον Τομπίας που εκπροσωπεί την Google. Εμάς θα μας ενδιαφέρει πάρα πολύ να μάθουμε γιατί η Google έχει αναπτύξει αναπτύξει Content ID για τη μουσική και το βίντεο και όχι για τις εικόνες, για τις φωτογραφίες. Γιατί δεν θα μπορούσε, για παράδειγμα, να δημιουργηθεί ένα Content ID και για τις φωτογραφίες και τις εικόνες. Και δεν έχουμε, δεν μπο, δεν έχουμε καμία δυνατότητα. Χρειαζόμαστε το νόμο για να μας προστατεύσει. Γιατί στα μέλη μας ε, συγκαταλέγονται και πολύ μικρές επιχειρήσεις, ατομικές επιχειρήσεις, για παράδειγμα οι οποίες χρειάζονται την προστασία του νόμου. Εμείς επιπλέον πιστεύουμε ότι ε, στην περίπτωση των εικόνων η οδηγία δεν πάει αρκετά μακριά, εκεί που θα θέλαμε εμείς. Γιατί δεν κλείνει διάφορες, διάφορους βρόχους, διάφορες, ε, ε, διάφορα κενά. Το άρθρο 13 αναφέρει μόνο το περιεχόμενο το οποίο αποθηκεύεται από την διαδικτυακή υπηρεσία. Και υπάρχει και αυτή η αιτιολογική σκέψη 33 όπου εξαιρούνται οι υπερσύνδεσμοι. Και όπως είπα υπάρχει διαφορά μεταξύ των συνδέσμων. Υπάρχουν σύνδεσμοι οι οποίοι καταλήγουν σε ένα συγκεκριμένο περιεχόμενο. Αυτό κάνουν ε, οι μηχανές αναζήτησης. Σου δείχνουν δηλαδή ότι πρέπει να πας σε εκείνη την κατεύθυνση, πατάς το link και πηγαίνεις στην ιστοσελίδα. Στην περίπτωση του, της εικόνας, όταν αυτές καδράρονται, το ε, link ταυτίζεται με την εικόνα. Αυτό είναι, είναι πάρα πολύ σημαντικό θα σας δώσω κάποια παραδείγματα για να εξηγήσω τι εννοώ. Εδώ βλέπετε αυτή την εικόνα. Έχει την άδεια ο Garden για 5,85 ευρώ. Κάποιο από τα μέλη μας παραχώρησε αυτή την άδεια στο Guardian. Βλέπετε εδώ ότι υπάρχει ένα σύστημα διαχείρισης περιεχομένου του Guardian. Η άδεια επιτρέψει τον πελάτη, εν προκειμένου τον Guardian, να ε, ε, επιτρέψει στους χρήστες να μεγεθύνουν την εικόνα αυτή. Εντάσσεται αυτή, αυτή η δυνατότητα στην άδεια που έχει παραχωρηθεί από το μέλος μας στον Guardian. Εδώ πατάς δεξιά πάνω και βλέπεις μια πολύ ωραία λεοπάρδαλη στο χιόνι. Αυτή η εικόνα λοιπόν είναι καδραρισμένη. Για, για το χρήστη το ίδιο πράγμα είναι. Ίσα ίσα η δεύτερη ε, εικόνα είναι και πιο όμορφη. Από τεχνολογική απόψεω όμω είναι διαφορετικό πράγμα. Η, ο, Guardian πλήρωσε 5,85 ευρώ στην, για την άδεια αυτή. Εντάξει, δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. Για ποιον λόγο όμω ε, η, η οδηγία δεν διακρίνει μεταξύ αποθηκευμένου και καθαρισμένου περιεχομένου. Εδώ βλέπετε ένα Google search ε, για, για εικόνα. Βλέπετε ότι υπάρχουν τρεις σελίδες όπου χρησιμοποιείται η ε, ε εν λόγω εικόνα. Στη γενική μηχανή αναζήτησης μπορείς μάλιστα να, να κάνεις και αναζήτηση για παρόμοιες εικόνες, οπότε δεν χρειάζεται καθόλου να πάει κανείς στην, στον φορέα που κατέχει τα δικαιώματα αυτής της εικόνας. Εδώ ε, βλέπετε μια οπτική εικόνα στο image search της Google, και βλέπετε ότι η εικόνα αυτή έχει αντιγραφεί σε μια σειρά από άλλες ιστοσελίδες. Βλέπουμε εδώ ένα άλλο παράδειγμα ενός άλλου μέλου μας για να σας δείξω ότι δεν υπάρχει διαφορά μεταξύ των αποθηκευμένων και των καδραρισμένων εικόνων. Βλέπετε εδώ ότι ε, υπάρχουν παράνομα αντίγραφα εικόνων των, των μελών μας και θα ήθελα να σας δώσω και ένα τελευταίο παράδειγμα, γιατί σχετίζεται με αυτό το κομμάτι της οδηγίας που αφορά, για παράδειγμα, ε, περίπου τον, το, τον, το διαμοιρασμό των εισόδων, των κερδών, για το κεφάλαιο 3 μήλο. Οι φωτογράφοι λαμβάνουν κάθε μήνα μια έκθεση για την χρήση των εικόνων τους. Αυτή την εικόνα, για παράδειγμα, ε, την, την, είχε, την είχε δώσει το AT Photos, Photostock στο Bing και εδώ ξαφνικά ο φωτογράφος αναφέρει ότι στην έκθεσή σας μου λέτε ότι ε, έχει χρησιμοποιηθεί η εικόνα μου μόνο δύο φορές. Εγώ όμως τη βρίσκω 242 φορές στο ίντερνετ. Το ότι αν είναι αποθηκευμένη ή καδραρισμένη η εικόνα αυτή δεν έχει σημασία. Γιατί δόθηκε, πουλήθηκε μία φορά η, η φωτογραφία αυτή ε, στην Bing, από εκεί και πέρα αντιγράφηκε 140 φορές και η, το πρακτορείο στο οποίο ανήκει η φωτογραφία αυτή δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Γιατί πληρώθηκε μόνο μία φορά, αλλά χρησιμοποιήθηκε δεκάδες φορές η φωτογραφία τη. Γι' αυτό χρειαζόμαστε τον νόμο για να μας προστατεύσει. Αυτό που έχει προταθεί είναι μια, ένα καλό πρώτο βήμα. Εμείς θέλουμε τη συνεργασία, αλλά θεωρούμε ότι δεν πηγαίνει αρκετά μακριά, γιατί δεν έχει κλείσει το, ε, το κενό αυτό του framing, του καδραρίσματος των φωτογραφιών. Κάτι που αφορά το 85% των εικόνων ε, των μελών μας. Ευχαριστώ πολύ. Αν ε, μας το επιτρέπουν οι συνάδελφοι και η Κομισιόν θέλει να κάνει μια δήλωση. Εν συντομία, σας παρακαλώ. Τρία-τέσσερα λεπτά. Η Κομισιόν δεν ε, ζήτησε συγκεκριμένα να κάνει δήλωση, αλλά ήθελε να ακούσει τις διαφορές απόψεις. Και νομίζω ότι αυτό που είναι σημαντικό να έχουμε κατά νου οι βουλευτές που ακούνε όλες αυτές τις πληροφορίες είναι η πραγματικότητα που περιγράψατε που περιγράψαν οι προσκεκλημένοι. Η Κομισιόν δεν θέλει να βάλει επιτέπτως μέτα κατά των πλατφόρμων ή κατά των καταναλωτών ή κατά των θεμελιωδών δικαιωμάτων ή κατά του ηλεκτρονικού εμπορίου. Βρίσκονται όλα αυτά στο επίκεντρο αυτό που κάνει η Κομισιόν, όμως η Κομισιόν και το Σώμα των Επιτρόπων ομόφωνα αποφάσισε ότι χρειάζεται ανάγκη παρέμβασης για να αυξηθεί η συνεργασία μεταξύ των μερών προκειμένου να διασφαλίσουμε ότι υπάρχει ένα μερίδιο της αγοράς για όλους ιδίω όταν βασίζεται στην εμπορική διανομή περιεχομένου που ανήκει σε κάποιον άλλον. Και αυτή είναι η ουσία της παρέμβασης ε, στο άρθρο 13. Άκουσα πόσο συγχυσμένη ήταν η τελευταία ομιλήτρια που θα ήθελε η Κομισιόν να πάει παραπέρα από τα προτινόμενα μέτρα στο άρθρο 13 και όλοι ξέρουμε πόσο δύσκολη είναι η συζήτηση για τα hyperlinks, για τους υπερσυνδέσμους. Όμως ε, νομίζω ότι ήταν ένα θέμα που εξήγησε πολύ καλά σε ό,τι αφορά τη χρήση των εικόνων ε, online με τεχνικές ε, όπως είναι ε, το να μπαίνουν σε κάδρο και ουσιαστικά αφαιρεί από τους φωτογράφους ε, να έχουν κάποια έσοδα από τις φωτογραφίες που βγάζεις. Νομίζω ότι χρειάζεται πολύς χρόνος για να πάρεις ε, μια καλή φωτογραφία μιας λοπάρδαλης με μπλεμάτια. Απλώς θα ήθελα να επαναλάβω λοιπόν ότι εδώ δεν δίνουμε μια μάχη κατά κάποιων συγκεκριμένων, αλλά γίνεται ουσιαστικά σύμφωνα με τη Χάρτα των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων και την Οδηγία Ηλεκτρονικού Εμπορίου και προκειμένου να έχουμε δικαιοσύνη στο επιγραμμικό εμπόριο, στην επιγραμμική αγορά και θα πρέπει φυσικά να συνεχίσουμε να προστατεύουμε τα δικαιώματα του δημιουργού. Ακόμη και αν δεν ζήτησα το λόγο και πάλι σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Τώρα έχουμε δύο λεπτά για ερωτήσεις και απαντήσεις. Κυρία Ρέντα. Έχω μια ερώτηση για τον κύριο Ρέινα. Αναφερθήκατε σε μηχανισμούς προσφυγής ε, και αν η πλατφόρμα λέει στους όρους χρήσης ε, δεχόμαστε απλώς αδειοδοτημένο περιεχόμενο. Και μια ακόμη ερώτηση σε εσάς και στην Κομισιόν η πρόταση δεν αναφέρεται σε παραβίαση του δικαιώματος του δημιουργού πουθενά λέει ότι οι πλατφόρμες ε, που έχουν πάρα πολλά έργα φορτωμένα θα πρέπει να έχουν αυτές τις τεχνολογίες αναγνώριση περιεχομένου όμως, τι γίνεται αν δεν υπάρχει κάποια παραβίαση copyright στη Wikipedia, παίρνοντα χάρη, όπου όλο το περιεχόμενο copyright καλύπτεται από μια άδεια θα πρέπει και αυτοί να έπρεπε να υιοθετήσουν τεχνολογίε αναγνώριση περιεχομένου ή θα πρέπει να κάνουν κάποιε συμφωνίες άδειαση με τους κατόχους των δικαιωμάτων ακόμη και αν δεν υπάρχει παραβίαση σε ό,τι φορά το δικαίωμα του δημιουργού, παράβαση ό,τι το δικαίωμα του δημιουργού. Ευχαριστώ πολύ. Δεν βλέπω να ζητά άλλο το λόγο. Ποιο θα ήθελε να απαντήσει στην κυρία Ρέντα. Αν κατάλαβα την ερώτησή σας καλά, μόνο οι πλατφόρμες, οι πλατφόρμες μόνο ε, περιεχόμενο το οποίο είναι αδειοδοτημένο θα μπορούν να χρησιμοποιούν. Τώρα αν ε, χρησιμοποιείται μία εικόνα και στο βάθος υπάρχει μουσική για ένα εορτασμό σαν παράδειγμα σε αυτή την περίπτωση το περιεχόμενο μπορεί να χρησιμοποιηθεί πολλαπλά και οι μηχανισμοί οι οποίοι ε, χρησιμοποιούνται σήμερα ελπίζουμε να συνεχίσουν να χρησιμοποιούνται στο μέλλον και το αν μπορείς να χρησιμοποιήσεις σωστά το περιεχόμενο εξαρτάται περισσότερο όχι από τους όρους με τους οποίους το έχει στη διάθεσή σου, αλλά από τον τρόπο με τον οποίο θα ε, χρησιμοποιήσεις τους όρους αυτούς. Και υπάρχει υποχρέωση επίσης από τα κράτη-μέλη να υιοθετήσουν και να εφαρμόσουν έναν μηχανισμό παραπώνων αναφορών αποζημίωσης και πώς αυτό λοιπόν θα ε, εφαρμοστεί από τα κράτη-μέλη θα πρέπει να έχουν μια υπηρεσία σαν παράδειγμα η οποία να δέχεται την ε, αναφορές παραπώνων για την χρήση του συστήματος. Εν πάση δεν ήμουν ασαφής. Η κυρία Κομοδίνη θέλει να θέσει μια ερώτηση. Χωρίς μικρόφωνο. Έχω πολλές ερωτήσεις, μία όμως θα κάνω. Νομίζω ότι η ερώτησή μου the meetings with different Λοιπόν, το θέμα είναι τον τρόπο με τον, για τον τρόπο που συνεργάζονται οι εμπλεκόμενοι, δηλαδή οι καλλιτέχνες, εκτελεστές, συνθέτες, τυχουργοί, μια ολόκληρη, αν θέλετε, αλυσίδα ανθρώπων που παρέχουν αξία. Το πρόβλημα είναι ότι όλοι, το παράπονο είναι ότι όλοι πληρώνονται, αλλά δεν πληρώνονται αρκετά. Μπορείτε να μας δώσετε ε, κατάλογο ε, περιεχομένου το οποίο κατεβάζετε και ε, για το οποίο υπάρχει μια κάποια κατανομή εσόδων. Γιατί από ό,τι καταλαβαίνω μέχρι τώρα αυτό διαφέρει. Αν αρχίσει ας πούμε το παιδί μου 9 ετών να τραγουδά και το περιεχόμενο μέσω ενός φίλου του κυκλοφορεί στο διαδίκτυο, ενώ κάποιος άλλος κατεβάζει ε, σε επίπεδο ε, επίσημο στα πλαίσια μίας από τις αναγνωρισμένες πλατφόρμες ένα αναγνωρισμένο περιεχόμενο. Γι' αυτό λοιπόν θα ήθελα να μας δώσετε τον πλήρη κατάλογο του περιεχομένου για τον οποίο θα υπάρχει ήδη κατανομή εσόδων. Δεν έχω τον κατάλογο αυτό, πρέπει να ρωτήσω τα μέλη μου, αλλά παρόλα αυτά αν μια βιντεοσκόπηση σαν παράδειγμα κατεβαστεί και ταυτόχρονα χρησιμοποιηθεί, αυτό είναι κάτι το οποίο καταμετράται μεν από τη μία, αλλά τι είναι αυτό το οποίο προκαλεί να ξεκινήσει η διαδικασία αποζημίωσης ή πληρωμής είναι κάτι στο οποίο δεν μπορώ να απαντήσω και δεν έχω κάποιον να με βοηθήσει για να δώσω απάντηση σε αυτό. Καλώς. Μας έδωσαν λίγα λεπτά περισσότερα οι διευμηνείς. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέλει ξανά το λόγο. για να απαντήσω ή να προσπαθήσω να δώσω μια απάντηση στην ερώτηση την οποία έθεσε η κυρία Ρέντα σχετικά με το είδος του περιεχομένου το οποίο κατεβάζεται και καλύπτεται από το άρθρο 13. Είναι κάτι που έχουμε συζητήσει ήδη διμερώς με την κυρία Ρέντα. Η ερώτηση είναι τι συμβαίνει στην περίπτωση που υπάρχουν πλατφόρμες που αποθηκεύουν περιεχόμενο το οποίο το κάνουν με άδεια του ε, παραγωγού. σε σχέση με τις αδειοδοτήσεις τύπου CCC, Creative Common License, CCL, συγγνώμη. Ίσως αυτό είναι ένα θέμα λοιπόν το οποίο πρέπει να διευκρινιστεί. Πρέπει να αντιμετωπιστεί το θέμα για το οποίο, σύμφωνα με το οποίο το περιεχόμενο και η αντιγραφή του περιεχομένου γίνεται χωρίς την εμπλοκή των παραγωγών, των κατόχων του δικαιωμάτων, των δικαιωμάτων κτλ. <coughs> Τίθεται θέμα εδώ με την ερμηνεία του άρθρου 13 δηλαδή δεν αφορά το θέμα πλατφόρμες οι οποίες φιλοξενούν περιεχόμενο το οποίο τους έχει δοθεί και αποθηκεύεται με τη σύμφωνη γνώμη του δημιουργού ή του κατόχου του δικαιώματος. Πάνω σε αυτό λοιπόν τίθενται ερωτήσεις όπως η Wikipedia αν περιλαμβάνεται ή εξαιρείται και γι' αυτό θα ήθελα να αναφερθώ στην αιτιολογική στο 37. Mrs. Comodini, who is the report... Τώρα η κυρία Κομοντίνη είναι η συγγήτρια για την πρόταση αυτή να κάνει τις καταληκτικές της παρατηρήσεις. Ευχαριστώ. Καταρχήν, θέλω να ευχαριστήσω όλους τους ε, ομιλητές που παρευρέθησαν εδώ σήμερα σε αυτή τη δημόσια κρόση. Νομίζω ότι ήταν ε, ιδιαίτερα χρήσιμη η συζήτηση. Κάτι που ανακάλυψα είναι ότι πολύ συχνά υπάρχει και παραπληροφόρηση ή ουσιαστικά θεωρούμε ότι γνωρίζουμε κάποια πράγματα σε ό,τι αφορά την προστασία των δικαιωμάτων δημιουργού και γι' αυτό θα ήθελα να πω ότι τους ευχαριστώ πολύ που παρευρέθησαν εδώ και για την ε, τις απαντήσεις που έδωσαν στις ερωτήσεις μας. Φυσικά η μεταρρύθμιση του δικαιώματος του δημιουργού είναι στα χέρια της Επιτροπής μας μόνο τους τελευταίους δύο μήνες. Όμως ε, έχουμε δουλέψει σκληρά και έχουμε συνεδριάσει πολλές φορές τους τελευταίους δύο μήνες για να βρούμε τις υποκείμενες ανησυχίες όλων των ενδιαφερομένων μερών. Εγώ θα συνεχίσω προς αυτή την οδό και καλό όλους όσους θέλουν να συζητήσουν περαιτέρω τα θέματα αυτά να έρθουν σε επαφή μαζί μου έτσι ώστε να μπορέσουμε να καταλήξουμε με μεταρρύθμιση του copyright που να αντικατοπτρίζει τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε σήμερα εντός ε, ε, του ψηφιακού τρόπου ζωή των πολιτών μα και για να διασφαλίσουμε ότι προστατεύονται τα δικαιώματα του δημιουργού και σε αναλογικό και σε ψηφιακό επίπεδο. Και κλείνω γιατί δεν θέλω να υπερβώ το χρόνο. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Να ευχαριστήσω και εγώ, όπως και η κυρία Κομοντίνη, τους ε, προσκεκλημένους μας που παρευρέθησαν στην ακρόαση αυτή να σας ευχηθώ καλή όρεξη.